Right, uh, welcome uh, we have an Καλώς ορίσατε. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Επίτροπο. Άργησε λίγα λεπτά, οπότε θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Επίτροπο, ο οποίος θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Πρόκειται για ένα μέρος του διαπνομένου διαλόγου. Ο κύριος Μπαρνιέ θα μας παρουσιάσει τις ε, προτάσεις ε, που θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή του επόμενους μήνες που αφορούν την εσωτερική αγορά και τις ε, διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρα. Σας χαιρετώ όλους και όλες. Συγγνώμη διότι καθυστέρησα λίγα λεπτά. Αλλά σήμερα το πρωί είχαμε την ε, συνάντηση των Επιτρόπων και μιλήσαμε για τη σημαντική πρόταση του συναδέλφου μου, του Καρέλ Ντεγκούχ, για τις παγκόσμιες αγορές και τους κανόνες αμοιβιότητες και γι' αυτό ίσως εξηγεί κάπως την καθυστέρηση. Ήμουν όπως και πολλοί από εσά την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και στην ώρα των ερωτήσεων στην οποία συμμετείχα για την ανταγωνιστικότητα, ή από τους συναδέλφους σας μου έκαναν ερωτήσεις για το θέμα της σημασίας των έργων υποδομής ε, στην ενιαία εσωτερική αγορά. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τις κατάλληλες βάσεις στην οικονομία μας στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και πάντα σκέφτομαι αυτή τα θεμέλια, τη βάση την οποία θα πρέπει σιγά σιγά να οικοδομήσουμε με μεγάλη υπομονή, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία μας να έχει την κατάλληλη βάση και να γίνει ανταγωνιστική και αηφόρος. Και να μην χτίζουμε σε κινούμενη άμμο, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν στα πλαίσια ή της αυτορύθμισης ή της έλλειψης οποιοδήποτε ρύθμισης και κανονισμού που είδαμε ότι ήταν ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε. Ό,τι κάνουμε μαζί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ και δύο χρόνια, συνίσταται συγκεκριμένα στο να δημιουργήσει υγιείς και σταθερές βάσεις διαφάνειας, ηθικής και ευθύνης ότι πολλές φορές η ηθική είδαμε ότι είχε εξαφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια ή να θέσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην πραγματική υπηρεσία της οικονομίας. Πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και στις προσδοκίες των πολιτών, πολλοί από τους οποίους υποφέρουν. Γι' αυτό, όπως μας ζήτησε το G20, πρέπει να θέσουμε το κατάλληλο πλαίσιο και η δουλειά η οποία γίνεται για τη διακυβέρνηση, για τη διαφάνεια και για τη ρύθμιση να γίνει εκ στην Ευρώπη όπως το κάνουμε πάρα πολύ ενεργά καθώς και στα άλλα μέρη του κόσμου, πράγμα το οποίο εξηγεί τον χρόνο τον οποίο μαλώνω εγώ στην Ουάσιγκτον σε τακτά διαστήματα και στο Τόκιο παρομοίως. Πρόκειται μόνο βεβαίως για ένα κεφάλαιο των όσων πρέπει να κάνουμε. Είναι το πρώτο κεφάλαιο. Δηλαδή, να ξαναδημιουργήσουμε πάλι υγιείς και σταθερές βάσεις, ένα σταθερό θεμέλιο για να μπορέσουμε να ε, κάνουμε την κατάλληλη εποπτεία της χρηματοπιστωτικής οικονομίας. Κάποιος άλλος, άλλου είδους επίσης πιο δυναμική ρύθμιση την οποία θα πρέπει να κάνουμε ενεργώντας εκ των προτέρων είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε με το shadow banking από κοινού. Με την προστασία των καταναλωτών και με τις διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις τράπεζες για να μπορέσουν να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ για όσους δεν είναι βουλευτές, για τους παρόντες που είναι ενδεχομένως οι δημοσιογράφοι για να καταλάβουν τι γίνεται και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το G20 ότι αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση πάρα πολλέ προτάσεις με την πολύ επικοδομητική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή το κείμενο το οποίο εσείς ε, ε, υιοθετήσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε έτοιμοι επίσης να υιοθετήσετε το κείμενο για τα παράγωγα του συναδέλφου σας, του κυρίου Λάγκεν, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στα πλαίσια αυτής των εργασιών πρέπει να πω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Κάτι το οποίο μπορέσαμε να κάνουμε, γι' αυτό το στα πλαίσια συνεργασία για αυτά τα θέματα θα πρέπει να το κάνουμε και για τις οδηγίες CDR και MIF. Ο κύριος ε, Καράς ασχολείται ενεργά με πάρα πολύ ε, με τα θέματα αυτά του CDR4 και επίσης θα ήθελα να πω ότι κανένας δεν θέλει να θέσει ένα αμφιβόλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, το οποίο θα θέσουμε για τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Για το ΜΥΦ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή Μάρκους Φέρμπερ. Η παρούσα ΜΥΦ θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα βήματα των ε, εναλλακτικών διαπραγματεύσεων οι οποίες γίνονται για τις ε, διαπραγματεύσεις υψηλής συγνότητας. Επίσης θα πρέπει στα πλαίσια της συνεργασίας να κάνουμε κάτι για τις καταχρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην αγορά ώστε να μπορέσουμε να καταστήλουμε οποιαδήποτε κατάχρηση υπάρχει σε σχέση με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέτρα που υπάρχουν μεταξύ ιδιωτών με κυρώσεις σαφείς και αξιόπιστες. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η οίκη αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντομενιτσί για την αποφασιστικότητά του. Επίσης, στα πλαίσια των εγγύσεων που αφορά τι καταθέσει. Θα ήθελα να πω ότι έκανε εξαιρετική εργασία ο εισηγητή σα, ο κύριο Πίτερ Σίμον. Και από την δική σας απόφαση θα κάνουμε στα πλαίσια της Δανικής ε, Προεδρίας το θέμα αυτό ώστε να μπορέσουμε με επικοδομητικό τρόπο να προχωρήσουμε σύντομα και, στην, ε, και να συμφωνήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία Omnibus 2 με τον Burkhard Balz και όλους σας και εγώ θέλω να μπορέσουν οι ασφαλιστές να προτείνουν πάρα πολύ καλές εγγυήσεις στις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και τελικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι και εμείς επίσης τον προηγούμενο Οκτώβριο υποβάλαμε προτάσεις για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, κυρίως τα 20 ε, εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επίσης θα πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα με το διαβατήριο για τις ε, εταιρείε του επιχειρηματικού κεφαλαίου με εισηγητή τον κύριο Λαμπέρ και τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις με εισηγήτρια την κυρία Οκονή. Επίσης, είμαστε σε συνεργασία με την Επιτροπή Τζούρι και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και τη συμφωνία στο πακέτο υπεύθυνε επιχειρήσεις και ζητήσαμε ε, καθώς και στη, να ασχοληθούμε με τον θέα των νέων οδηγιών που αφορούν την εξορρυκτική βιομηχανία και, ε, και την ε, υλοτομία. Εκθέσεις καθώς και την οδηγία για τη διαφάνεια πρόκειται για τις εκθέσεις Clinch και Πίτι Canyon. Όπως σας είπα, Όλα αυτά τα κάνουμε προσπαθώντας να μάθουμε και από την κρίση. Δεν ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε να προχωρήσουμε ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και όπως σας είπα την πρώτη μέρα της ακρόασης, καμία χρηματοπιστωτική αγορά και κανένα προϊόν και κανένας φορέας δεν θα πρέπει να αποφεύγει την ε, ρύθμιση και την εποπτεία. Οι προτάσεις λοιπόν που έχουμε μπροστά μας, που περιμένουν όπως και εσείς η κυρία Φερέιρα και ο κύριος Χόκμαρκ, είναι προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης και την επίλυση της κρίσης. Το σχέδιο αυτό θα το παρουσιάσουμε σε έφθετο χρόνο. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση εσωτερικής διαβούλευσης και η διαβούλευση αυτή ίσως θα επεκταθεί και σε διάφορους υπευθύνους και εμπλεκόμενους stakeholders, κυρίως όσον αφορά το θέμα το πολύ ευαίσθητο του bail-in και το σύνολο των μέτρων που θα υιοθετήσουμε, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει και το timing να είναι καλό και το σύνολο των μέτρων ώστε να ε, μπορέσουμε με αυτό το στοχευμένο τρόπο τις επόμενες εβδομάδες να παρουσιάσουμε το κατάλληλο κείμενο. Επίσης, ένας άλλος τομέας που ενδιαφέρει πολλούς από εσά και δικαίως, δεδομένου ότι μιλούμε για γενικότερη δημόσια ρύθμιση, είναι το shadow banking. Έχει αρχίσει η διαβούλευση για το θέμα αυτό και ξέρουμε ότι το θέμα αυτό των μη τραπεζικών πιστώσεων που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή έχει άμεση ή έμεση σχέση με το τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες και σε διεθνές επίπεδο και το Συμβούλιο ε, Χρηματοπιστωτική σταθερότητος και το G20 θέλουν να κάνουν συστάσεις επί αυτού του θέματος. Θα οργανώσουμε για το θέμα αυτό μία διάσκεψη στις 27 Απριλίου που θα αφορά το shadow banking, τους κανόνες για την τράπεζα και θα ήθελα και εσείς να μπορέσετε να συμμετάσχετε. Ο τρίτος άξονας. Ένα άλλο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με το οποίο θα ασχοληθώ φέτος είναι το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα εμπιστοσύνη και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οικοδομήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών και των τραπεζών. Υπάρχουν πάρα πολλά τοξικά προϊόντα, υπάρχουν προϊόντα τραπεζικά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στι ανάγκε. Πολλά είναι πάρα πολύ δαναπανηρά και η πρόσβαση στην σωστή ενημέρωση δεν είναι πάντα σωστή. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει και πάλι εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις τράπεζες, θα πρέπει να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των καταναλωτών προς τον κόσμο των τραπεζών. Επίσης, πέρσι αρχίσαμε να εργαζόμαστε σε θέματα ε, εν υποθήκων δανείων με την εισήγηση του, κυρίου, με την, του κυρίου Σάντζετ Πρεσέδο και θα παρουσιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες για τα πρίψ, τα ε, προϊόντα επενδύσεων ιδιωτικών. Πρόκειται εδώ για ποσά της τάξεως των 11 ε, δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2009 και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος και ποιος είναι ο κίνδυνος που ενέχουν όλα αυτά τα προϊόντα. Επίσης υπάρχουν ε, τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κυρία Πέρες που αφορούν τα διάφορα επενδυτικά κεφάλαια, τα δομημένα προϊόντα και τα λοιπά και, τα λοιπά και κάποια προϊόντα που αφορούν τις ε, ασφάλειες ζωής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία καταλήγουμε, τα μαθήματα που μαθαίνουμε από την απάτη Μάντοφ και από τις δυσλειτουργίες του όλου τραπεζικού συστήματος και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε του καταθέτε. Όσον αφορά τις, την ε, διαμεσολάβηση σε θέματα ασφαλιών, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε επίσης και εκεί κάτι. Επίσης θα συνεχίσουμε να, συνε... να ασχολούμαι με μια οδηγία που πολλές φορές έχει προκαλέσει επικρίσεις, που είναι το θέμα των συντάξεων, συνταξιοδοτικών ταμείων, πράγμα που πολλές φορές έχει ανησυχήσει τους πάντες και πολλές φορές στον τύπο δεν εμφανίζεται η σωστή εικόνα. Η πρόθεσή μας δεν είναι να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες ρεστότητες στα, για τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και να είμαστε προσεκτικοί ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία προτείνει κάθε συνταξιδοτικό ταμείο. Επίσης, θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο για τις προθέσεις μου όσον αφορά αυτό το θέμα της χρηματοδότησης μακροπρόθεσμα, δεδομένου τα συνταξιοδοτικά ε, ταμεία είναι σημαντικά για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Βεβαίω, αυτό είναι ο ρόλο των τραπεζών, αλλά εκείνο το οποίο με απασχολεί εμένα είναι οι συνέπειες ή ο αντίκτυπο όλων αυτών των κανονισμών και διακανονισμών που ζητά το G20 όσον αφορά την χρηματοδότηση οικονομίας μακροπρόθεσμα. Και θα ήθελα να αρχίσει συζήτηση σημαντική από αυτού του θέματος με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και ενεχόμενους συναδέλφους, τον κύριο Όλι Ρέν και τον κύριο Ταγιάννη, προτείνοντας μία πράσινη βίβλο για την χρηματοδότηση της οικονομίας και τη χρηματοδότηση την ε, μακροπρόθεσμη τους επόμενους μήνες. Το τελευταίο σημαντικό θέμα αφορά τους καταναλωτές. διαφάνεια όσον αφορά τα, ε, το κόστος των τραπεζών, τα ποσά που χρεώνουν οι τράπεζες, πράγμα το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε καταναλωτή να κάνει σύγκριση και γι' αυτό μεταξύ όλων των δαπανών και γι' αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα ε, σαφής η κατάσταση για τους καταναλωτές. Το switching επίσης είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε και τον Ιούλιο του 2011 το μήνυμα το οποίο στείλαμε ήταν αρκετά σαφές, πράγμα το οποίο όπως τη βλέπουμε δεν είναι επαρκές, γι' αυτό θα εργαστούμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μία νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό. Και εδώ αναφέρομαι στην έκθεση πρωτοβουλία του συναδέλφου σας κυρίου Κλίτεν. Κυρίες και κύριοι, τελείωσα προς το παρόν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ίσως δυο λόγια ακόμη για ένα δομικό πρόβλημα. Απαντώντας τον κύριο Λάμπερτ, εδώ και κάποιους μήνες είχα αναλάβει την εξής δέσμευση για το θέμα αυτό. Πρέπει να αναλώσουμε χρόνο και να εργαστούμε σύντομα και σοβαρά για το θέμα του διαχωρισμού των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, επιλέγοντας σωστά τα άτομα τα οποία μελετούν αυτά τα θέματα ε, υπάρχει ομάδα εργασίας της οποίας προεδρεύει ο πρώην συνάδελφος Βερλικάνεν, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της, Τράπεζας της Φιλανδίας και γύρω στα 10 άτομα εργάζονται για αυτά, γύρω από αυτά τα θέματα και βλέπουν τι γίνεται και με την Volker Rule και με το τι ακριβώς γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία. Θέλω να, γίνουν, να έχουμε πληροφορίες πλήρεις, ανεξάρτητες, και νομίζω κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών αυτής της ομάδας που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο θα πρέπει να υπάρξει και διαβούλευση της δικής σας Επιτροπής ώστε να μπορέσετε κι εσείς να γνωμοδοτήσετε πάνω σε αυτά τα οποία θα έχει κάνει η ομάδα Λικάνεν. Βεβαίως τίποτα δεν σας εμποδίζει και εσείς να προσθέσετε τις δικές σας ιδέες όσον αφορά τον χωρισμό των κινδύνων και το τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται λοιπόν και για ένα Άλλο θέμα, πολύ σημαντικό και από τις εργασίες τις οποίες θα καταλήξει η ομάδα Λικάνεν θα μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω προτάσεις. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank you very much. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη παρακαλώ να μου δώσουν ένα λεπτό. Ξέρετε ότι δεν κλέβω συχνά χρόνο όταν έχουμε εδώ επιτρόπους, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω πρώτα απ' όλα. Θα θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε στη συνειδρίαση για το banking, αλλά ξεχάστε να με καλέσετε ως κύριο μιλήτρια, ενώ είναι κάτι το οποίο γνωρίζω καλά και το έχω αποδείξει στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κανονίσουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι απλά είναι μια μικρή παράληψη αυτό εκ μέρου σα. Ε, είστε καλεσμένοι. Α, πολύ ωραία. Δεν βρίσκομαι στο πρόγραμμα, αλλά θα το... Στις 27 λοιπόν, πολύ καλά. Όσον αφορά το ζήτημα της μακροπροθέσμης χρηματοδότησης και των ε, τραπεζών, θα ήθελα να σας σχολιάσω ορισμένες ομιλίες. Σας διαβεβαιώ ότι θέλουμε μια, να κάνουμε μια αρχική έκθεση που θα αφορά την απόκριση και θα το συζητήσουμε μεταξύ συντονιστών σύντομα. Ε, μια έκθεση πρωτοβουλίας λοιπόν. Τώρα ορισμένα ζητήματα Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γνωρίζετε. Υπάρχουν πέντε νομοθετικές πράξεις, όχι όλες δικές σας, που μπορεί να φτάσουν σε στάδιο τριμερούς διαλόγου πριν το καλοκαίρι, όπως η οδηγία απαιτήσεων κεφαλαίου. Μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από ένα τριμερής διάλογοι και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα χρειαστεί να ορίσουμε προτεραιότητες. Δεν θα μπορέσουμε να τους διεκπαιρεώσουμε όλους. Ε, για παράδειγμα, την υλοποίηση των στατιστικών στοιχείων, που είναι αρκετά σημαντικό σημείο. Αν δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα, επειδή δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ο όγκος της νομοθεσίας είναι τόσο μεγάλος. Ε, δίνω τώρα το λόγο στον Πολ. Ναι. Για τις ερωτήσεις σας. Δεν έχω ερωτήσεις. Πάντα είναι πολύ ακριβής ο Επίτροπος. Απαντά εκ των προτέρων της ερωτήσεις μας. Αφού μου δίνετε το λόγο, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω στον Επίτροπο ότι δεν είναι επειδή έχουμε πολλούς φακέλους που δεν θα τους αντιμετωπίσουμε σωστά. Θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουμε εξίσου καλή εργασία όπως και οι δικές σας ομάδες. Έχουμε ένα πρόβλημα και το λέω δημοσίως εδώ το νέο κανονισμό για τη διερμηνία που ουσιαστικά παραλύει εν μέρη τις εργασίες μας. Εσείς φυσικά δεν εμπλέκεστε σε αυτό, αλλά σας εξηγώ κύριε Επίτροπε ότι αν μια μέρα οι συγητές, οι σκιώδεις αποφασίσουν να πάψουν να εργάζονται θα είναι διότι δεν θα μπορούν να εργάζονται σε μια κοινή γλώσσα. Η δημοκρατία σε αυτό το κοινοβούλιο είναι η πολυγλωσία. Η εργασία των διερμηνέων είναι αναγκαία. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να εργαστούμε και θεωρούμε τώρα ότι με αυτή την ανόητη πολιτική μείωση των δαπανών για τη διερμηνία δεν θα έχουμε πλέον ε, διερμηνία όταν θα συζητάμε για παράδειγμα κατεξουσιοδότηση πράξης που είναι σημαντικό ε, θέμα δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι αν δεν μπορούμε να εκφραστούμε τουλάχιστον σε δύο-τρεις γλώσσες ε, δεν αξίζει καν τον κόπο να κάνουμε τη δουλειά μας και σήμερα ήμουν σε συνεδρίαση για το Τούπακ και μετά από 7 χρόνια που είμαι βουλευτής υποχρεώθηκα να παίξω το χαρτί μου του συντονιστή ώστε να, μου, να έχω τις υπηρεσίες ενός δερμηνέα για ψιθύρισμα ο οποίος δεν μπορούσε να πάει στις καμπίνες για να μεταφράσει τα αγγλικά. Ε, δεν φταίτε εσείς φυσικά γι' αυτό, αλλά σας το λέω για να γνωρίζετε ότι δεν διευκολύνει το έργο μας κάτι τέτοιο και τα όργανα αυτού του κεφαλαίου, ε, τα μέλη αυτού του ε, κοινοβουλίου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα οι Εάν θέλουμε η δουλειά μας να γίνεται σωστά, θα πρέπει να μπορούμε να εκφραστούμε σωστά. Ωραία είναι να μιλάμε όλοι πάντα αγγλικά, αλλά δεν είναι σωστό. Αυτό ήθελα να σας πω κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Κατά τα άλλα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα δουλέψουμε σκληρά και θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο ύψος των όσων μας προτείνεται. Πιστεύω ότι επίσης είναι σημαντικό και το αναφέρω διότι στον τύπο οι δημοσιογράφοι το αναφέρουν ε, συχνά. Ήθελα να αναφέρω επίσης και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, θέλω να ξέρετε ότι όσοι εκφράζουν την άποψη αυτής της Επιτροπής είναι οι εκθέσεις που ψηφίστηκαν με πλειοψηφία και όσοι επιφορτίστηκαν με την παρουσίαση αυτών των εκθέσεων στους τριμερείς διαλόγους που αποτελούν την έκφραση της βούλησης της παρουσίας Επιτροπής. Πιστεύω ότι επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε οι τριμερείς διάλογοι να αποτελούν μια ευκαιρία επαναδιαπραγμάτευσης θέσης ε, μειονοτήτων του Κοινοβουλίου. Μου δώστε το λόγο. Σας ενθαρρύνω κύριε Επίτροπε. Α, μάλιστα για τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας ε, Πιστεύω ότι χάρη στο φίλο μας τον κύριο Ντομίνιτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα ταράξουν κάπως ε, τα ήρεμα νερά στα οποία πλέον ορισμένοι οργανισμοί επιστοληπτικής ικανότητας και ελπίζουμε ότι θα εκτιμήσετε τις προτάσεις μας αυτές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Je peux répondre comme ça, d'entre vous. Μπορώ να σας απαντήσω ε, απευθείας ε, δεν πρέπει να υπάρχει αμφισημία ούτε έλλειψη κατανόησης. Εγώ έχω ανάγκη σας ε, σε αυτή, την παρουσία σας σε αυτή τη συνειδρίαση της 27 Απριλίου για το Shadow Banking. Σας, έχω, σας έχει σταλεί μια επιστολή, θα φροντίσω να επαληθεύσω ότι έχει όντως σταλεί και αν χρειαστεί θα επαναλάβω, θα ξαναστείλω την ίδια επιστολή. Υπολογίζω σε εσά και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας. Υπολογίζω ότι θα συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, δημόσια συζήτηση για το shadow banking, για τη σκιώδη τραπεζικά συστήματα. Γνωρίζω ότι επιτελείται σημαντικό έργο. Ζητείτε πολλή δουλειά από τα μέλη αυτής της ε, Επιτροπής, ε, γνώσεις, ικανότητες, ε, ακρίβεια και σας ευχαριστώ εσάς ε, όσο και τους διερμηνείς. Δεν γίνεται να γίνουν όλα μαζί. Ε, μου λέτε εσείς ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Ε, εγώ προσπαθώ σε λιγότερο από δύο χρόνια με όλες μου τις ομάδες και το γραφείο και τη Γενική Διεύθυνση Ευχαριστώ πολύ για τις ευχαριστήσεις και η κυρία Καλβίνο επίσης ήθελα να να, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της. Ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Ε, σίγουρα το BFID, οι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας, για τους οποίους μόλις μιλήσατε, καθώς και το διαβατήριο για τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτά είναι ορισμένα σημεία που θα θέλαμε να διεκπαιρεώσουμε χωρίς καθυστέρηση. Ε, στη συνέχεια, αν αποκτήσετε εσάς, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. ώστε να προσφέρετε μερικά χαμόγελα στην περιοχή μου υπάρχει μια έκφραση ε, στις Άλπεις ε, ε, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα για να κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο αναφέρει ο μιλητής στα γαλλικά ευχαριστώ κύριε Κωνσής για Δεν θέλω να σας να αναφερθώ στη διερμηνία για την οποία, την οποία χρειάζεστε. Υπάρχει ένα άλλο θέμα ε, στο πλαίσιο των ε, δραστηριοτήτων μου στην εσωτερική αγορά. Προσπαθούμε να επισπεύσουμε ένα θέμα που δεν θα μας απαλλάξει από τους διερμηνείς αλλά θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ μας, την ηλεκτρονική μετάφραση ώστε τα έγγραφα να μεταφράζονται με υψηλή ποιότητα ηλεκτρονικά και το μελετάμε αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Είναι δυνατός αυτός, αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν μια σωστή μετάφραση, να παρέχουν σωστή μετάφραση. Φυσικά η γραπτή μετάφραση είναι διαφορετική από την προφορική. Thank you very much. Um, I'll now move on. Ευχαριστούμε πολύ, επειδή πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ να είναι σύντομες οι ερωτήσεις για να μπορούν να είναι σύντομες και οι απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας. Πάντα με ευχαρίστηση. Σας δεχόμαστε για να καταλάβουμε πώς ε, διασυνδέονται με το Κοινοβούλιο οι δικές σας πρωτοβουλίες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Χαιρετίζω την ε, δική σας πρωτοβουλία για το shadow bankers, για τις μη ρυθμιζόμενες τράπεζες και την πρωτοβουλία σας να στήσουμε περισσότερο το bail-in να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τράπεζες. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά η ερώτησή μου αφορά. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εργασίες για να έχουμε μία νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα που αφορά τις τράπεζες. Διότι εμείς πρέπει να πω ότι είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Οι χώρες που ακόμη δεν μπορούν να προστρέξουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όλο και περισσότερο μεγάλο χρέος έχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί έναν, ε, έναν ε, φαύλο κύκλο. Αυτός ο οποίος πληρώνει όμως τα σπασμένα σε όλη αυτή την ερώτηση είναι ο κάθε φορολογούμενος. Πότε λοιπόν και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας θέσω αφορά την ε, ε, χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, που είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Με ποιο τρόπο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εισαγάγει κανόνες ώστε η, τα δάνεια που κάνει στις διάφορες εμπορικές τράπεζες, η κεντρική τράπεζα, να μπουν πραγματικά και να χρησιμεύσουν στην πραγματική οικονομία. Διότι αυτό το οποίο γίνεται είναι να διευκολύνονται οι τράπεζε, αλλά να μην υπάρχει ρευστό στην αγορά και κυρίως να υποφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρετε δύο σημεία. Θα απαντήσω κι εγώ με συντομία. Κυρία Φερέρα, αν δείτε την ενδεικτική, τον ενδεικτικό κατάλογο των δραστηριοτήτων μας όσον αφορά το shadow banking, βλέπετε ότι υπάρχουν ε, εργαλεία επενδύσεων σημαντικά. Ε, διαμεσοβαλαβητές ε, πιστώσεων, όλοι αυτοί οι οργανισμοί που παίζουν το ρόλο, αν θέλετε, των head funds που όμως δεν υπόκεινται καθόλου ή τουλάχιστον υπόκεινται μόνο εν μέρη στους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις. Θα αναφερθώ επίσης και στην τιτλοποίηση. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί αυτό το shadow banking που είναι 30-35% του τομέα αυξάνεται. Αυξάνεται. Διότι ένας μεγάλος αριθμός των ε, εργαλείων όπως κύριε Γκοζές το IFM και το MIFID θα πρέπει κανονικά αν υιοθετηθούν τα μέτρα που έχουμε προτείνει να οδηγήσουν στη μείωση του τομέα αυτού, στη μείωση του shadow banking. Γιατί, γιατί χάρη στις διαβουλεύσεις μας, χάρη στις εργασίες μας, θα πρέπει να εντοπίσουμε πού βρίσκονται τα αδύναμα σημεία και να τα καλύψουμε με νομοθετικά κείμενα. Αυτό ελπίζω το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον πριν το τέλος του έτους. Τώρα, μιλήσατε για την πραγματική οικονομία. Εγώ σας παρουσίασα τις προθέσεις μας όσον αφορά τις τομιακές ρυθμίσεις, κάθε αγορά, κάθε φορέα. Θέλουμε να έχουμε μία ευρύτερη εικόνα της χρηματοδότησης και να δώσουμε και κάποια κίνητρα, όπως παραδείγματος χάριν το διαβατήριο για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, όλα τα μέτρα για τις κοινωνικές ε, επιχειρήσεις. Όπως είχα πει και στην Επιτροπή πριν από λίγες ε, εβδομάδες, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε κι εσείς, να μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία και για τη χρηματοδότησή της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και γι' αυτό και μίλησα και με το ο Λιρέν, τον συναδελφό μου. Πριν από τέσσερις ή πέντε μήνες βρισκόμασταν σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Το διατραπεζικό σύστημα ήταν εντελώς μπλοκαρισμένο, δεν λειτουργούσε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έπαιξε το ρόλο της δίνοντας μια νέα όθηση στο διατραπεζικό σύστημα ελέγχοντας βεβαίως ότι τα χρήματα που τροφοδότησαν ε, την αγορά διοχετεύθηκαν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, ο τελικός αποδέκτης πρέπει να είναι η πραγματική οικονομία. Επαναλαμβάνω, είμαι σε στενή επικοινωνία με τον Όλυ Ρεν και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Ο Σφεν. Ναι, θα μιλήσω γερμανικά, έτσι ώστε ο Ζομπόλ να μην χρειάζεται μετάφραση και να κάνουμε και κάποιες εξοικονομήσεις όσον αφορά τα έξοδα διερμηνίας. Κύριε Επίτροπε, μιλήσαμε σήμερα και ψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή για το Omnibus 2. Όσον αφορά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, μιλήσαμε για τις υποχωρήσεις ε, στο ασφαλιστικό σύστημα, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις της κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μία ερώτηση. Η πρόταση όσον αφορά εγγύσεις για το ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει μία έκθεση πρωτοβουλίας, όπως ξέρετε, και το θέμα ξαφνικά χάθηκε. Η έκθεση δεν ξέρουμε τι απέγινε. Ανησυχώ λοιπόν και πραγματικά περιμένουμε όλοι κάποιες εγγύσεις, ένα σύστημα εγγύησεων. Δεύτερον, αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι πέρα από το σύστημα των εγγύσεων, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Και ενδεχομένως εδώ υπάρχουν προτάσεις από μέρους Επιτροπής. Μία πρόταση διαχείρισης κρίσης, θα έλεγα, για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πληρώσουν την ύφη οι τελικοί καταναλωτές, οι πελάτες τελικά των ασφαλιστικών εταιριών, αν θέλετε. Πώς μπορούμε να προτείνουμε ένα σύστημα εγγύσεων το οποίο να λειτουργεί. Ναι, βεβαίως μπορώ να απαντήσω. Πρόκειται για μια προσπάθεια όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων στον ασφαλιστικό τομέα. Αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει. Όπως ξέρετε, εδώ και τέσσερα χρόνια ασχολούμαστε με την διάσωση των τραπεζών. Εδώ και τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μία σειρά άτακτων, άτακτων και όχι οργανωμένων πτωχεύσεων στο τραπεζικό σύστημα. Και για να μην οδηγηθούμε σε ένα σύστημα όπου ο τελικός καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει, όπως είπατε, θελήσαμε να λυθούν κάποια μέτρα. Γιατί βεβαίως ο φορολογούμενος είναι αυτός που τελικά χρηματοδοτεί αυτού του είδους τις ε, καταστάσεις. Κύριε Γκίγκολτ, βεβαίως και πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών. Όπως ξέρετε, το 2010 υποβάλαμε μία λευκή βίβλο για το θέμα αυτό και οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν, θα έλεγα, καθυστερήσει, αναβληθεί, διότι είχαμε άλλες προτεραιότητες. Την οικονομική κρίση. Δεν φταίτε εσείς, βεβαίως. Αλλά και εσείς αυτή τη στιγμή έχετε καθυστερήσει στις εργασίες σας εξαιτίας της δικής μας καθυστέρησης. Τι να σας πω, είχαμε το G20 και τα μέτρα που έπρεπε επιγόντως να λυθούν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Θέλω να επωφεληθούμε από όλες τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα ε, αυτήν την εποχή για τις καταθέσεις και για τις επενδύσεις, αλλά η ανάλυση αυτή θα συνεχιστεί και το 2013. Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω ότι αυτή η οικονομική κρίση συμβαίνει παράλληλα με το Solvency 2. Ε, την ξέρετε την ιστορία. Τα κείμενα υπάρχουν, τα κείμενα είναι γνωστά και η Ευρωπαϊκή... Α, συγγνώμη, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Η Βίκη. Επίτροπε, χαίρομαι πολύ που Λοιπόν, θα κάνω τις ομάδες μία προς μία με τις πρώτες τους ερωτήσεις και μετά θα τις ομαδοποιήσω. Επίτροπε, χαίρομαι που σας ακούω να μιλάτε για τις επιπτώσεις της νομοθεσίας της μακροπρόθεσμης επενδύσεις ορισμένη από εμάς εδώ που έχουμε ζητήσει τις ωρευτικές επιπτώσεις για τις ακούσει συνέπειες εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα το πρωί στην άλλη μου επιτροπή βιομηχανίας και ενέργειας έγινε μια άλλη ψηφοφορία όπου κάθε όλοι υποστήριξαν ένα έγγραφο για τις επενδύσεις στην Ευρώπη και επισήμαναν την ανάγκη για ε, ε ουσιαστικά που θα βοηθήσουν στη δημιουργία υποδομής για επενδυτές όπως ασφαλιστές θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτό και ανησυχώ διότι η πράσινη βίβλος μπορεί να βγαίνει με τις καλύτερες προθέσεις αλλά μπορεί να μην είναι αρκετά γρήγορη για να προβλέψει ακούσεις συνέπειες. Είναι πολύ περίπλοκη νομοθεσία αυτή η οποία εισάγουμε. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να δράσουμε γρήγορα και να κάνουμε τροποποιήσεις στην νομοθεσία αν χρειαστεί. Είναι μεγάλη τύχη που εσείς και άλλοι καταφέρατε να αναλάβετε δράση για τη Φερεγγιότητα 2 την περασμένη εβδομάδα, αλλά αν είχε γίνει λίγες μέρες μετά από την ψηφοφορία ή λίγες μέρες πριν, ε, ορισμένοι επενδυτές σε υποδομές ε, είχαν εκφράσει τις ε, ανησυχίε του, τότε το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Η λιγες μερες πριν ορισμενοι επενδυτες σε υποδομες ειχαν εκφρασει τις ανησυχιες τους τοτε το προβλημα θα ηταν πολυ μεγαλυτερο η ερωτηση μου λοιπόν είναι πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι στα επόμενα χρόνια και τους επόμενου μήνε μπορούμε να αντιδράμε πιο γρήγορα στι ακούσεις συνέπειε ορισμένων από τι νομοθεσίε μα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο για το, χρηματοπιστωτική νομοθεσία γενικότερα. Euh, Ευχαριστώ που το αναφέρετε, Βίκυ. Όπως είπα προηγουμένως στην κυρία Φερέρα και στην εισαγωγή μου, αυτό το ζήτημα που με απασχολεί καθημερινά το να επιλέξουμε τις σωστές ρυθμίσεις για κάθε κείμενο, τη σωστή ισορροπία, όπως κάναμε από την αρχή, κύριε Φόρντ, για το ζήτημα των ε, ασφαλιών, ε, ε, για το Omnibus και το Solvency. Η τρίτη αυτή η ισορροπία στην οποία πρέπει να προσέχω είναι η διατλαντική ισορροπία δηλαδή ο παραλληλισμός των μέτρων που παίρνουμε εμείς για να οικοδομήσουμε ε, ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού πρώτα με τους Αμερικανούς γιατί 80% των συναλλαγών μας είναι διατλαντικές και προοδευτικά με τις υπολείπες περιοχές του κόσμου. Αυτή η εργασία για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, ε, κυρίως όσον αφορά τις ασφάλειες δεν έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εργασία για τον Omnibus ε, και τα υπόλοιπα κείμενα. Τα κείμενα που παρουσιάζουμε σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Φόρντ, ε, ε, φροντίζω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τηρώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί από τους αρχηγούς κρατών, του G20, και για σε οποίες δεσμεύσεις έχουμε συμφωνήσει όλοι. Για παράδειγμα, η πρόταση που κάναμε για τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα, ευελιξία στο εσωτερικό της ενία αγοράς για τις νέες επιχειρήσεις. Όπως το εργαλείο που προτείναμε για ένα πολύ σημαντικό τομέα της ε, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ε, στο MIFID αναζητήσαμε τα μέσα για να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να, να χρησιμοποιούν ένα σήμα σε πολλά κείμενα που αφορούν τη διαφάνεια. Έχουμε διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιορίζοντας τις λογιστικές υποχρεώσεις. Για αυτά τα πράγματα με ρημνώ τώρα εγώ. Θα ήθελα, τώρα που έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στη δουλειά μας σε αυτά τα κείμενα μαζί σας, θα ήθελα να σας θέσω την εξής ερώτηση για αυτή την πράσινη βίβλο με τον κύριο, που την συζητώ με τον κύριο Ρέν και τον κύριο Ταγιάννη. Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση ώστε να καταλήξουμε στα καλά προληπτικά, προορατικά μέτρα, δυναμικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Μου κάνετε νόημα κάτι δεν απαντήθηκε. Το ζήτημα μου είναι ότι αφού εγκριθούν τα κείμενα και ξέρω ότι κάνουμε πολλή δουλειά για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη σωστή διατύπωση των προτέρων, το ζήτημα είναι τι συμβαίνει όταν φτάνουμε σε στάδιο υλοποίηση ή ορισμένε φορέ όπω έχει συμβεί ήδη σε συζήτηση επίπεδου 2 και εκεί ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ακούσιες συνέπειες και εκεί αυτό το κοινοβούλιο και αυτή η επιτροπή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ακούμε την πραγματική οικονομία και όχι απλά την έγκριση της νομοθεσίας. Ότι ακούμε και τη ρεαλιστική πτυχή. Πιστεύω ότι είναι μια συνεχής εργασία, μια εργασία να εξελίξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό. Απλά να σας πω, όταν ήμουν υπουργό στη χώρα μου, Έλεγα ότι έδινα πολύ σημασία στην παρακολούθηση όσο και στην πρόβλεψη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στο Κοινοβούλιο και στην ε, Επιτροπή να παρακολουθούμε τα κείμενα. Αυτό γίνεται πολύ καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι μερικέ φορέ σε εθνικό. Το ίδιο και όσον αφορά τα μέτρα επίπεδου 2. Σε πολλά από αυτά τα κείμενα, κυρία Φόρντ, έχουμε ένα εργαλείο τη ρήτρα αναθεώρηση, επανεξέταση ε, στα περισσότερα από αυτά τα κείμενα έχουμε εισαγάγει μια τέτοια ρήτρα για να επιλύουμε προβλήματα, για να καταλήγουμε σε συμβιβασμού, η οποία χρησιμοποιείται αυτή η ρήτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των κειμένων. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί ιδιαίτερω. Okay, thank you. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο στι ε, ατομικέ ερωτήσει, ο Γιώργεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αρχικά, κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Από τη δική μου άποψη πολλά σημεία μπορώ να τα στηρίξω. Είναι βέβαιο ότι προχωράμε σε μια σαφή ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών που, την οποία εγώ επικροτώ ως εισηγητής για ε, το Financial Inclusion. Έχω να κάνω μερικά σχόλια. Στις 6 Μαρτίου η Κομισιόν δημοσίευσε μια σύντομη ανακοίνωση που παρουσίαζε τις αντιδράσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη σύσταση του περασμένου Ιουνίου. Ε, ακουγόταν σαν περιοδικό, σαν ε, έρευνα περιοδικού. Δέκα χώρες δεν απάντησαν καθόλου. Ορισμένες άλλες χώρες ε, λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να δράσουμε. Μια χώρα θεωρεί η Εθνική Τράπεζα έγραψε μια επιστολή βασικά η οποία λέει ότι οι... κλήθηκαν οι τράπεζες της χώρας να συμφωνήσουν στην ανακοίνωση της Κομισιόν, πολύ περίεργο πράγμα. Σε μια άλλη χώρα είπαν ότι τον Ιούνιο του 2010 είχαν υιοθετήσει νομοθεσία και ο πληθυσμός δεν την χρησιμοποίησε. Έτσι, συνεπώς, τον Απρίλιο του 2011 είχε ήδη καταργηθεί η νομοθεσία. Όλα αυτά ε, είναι σαν να προέρχονται από κάποιο ανέκδοτο. Αυτού του είδους ε, η ενθάρρυνση σε θελοντική δράση δεν βοηθάει. Χρειαζόμαστε δεσμευτική νομοθεσία. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι είναι πραγματικά απαραίτητο για εμάς να προχωρήσουμε προς δεσμευτική νομοθεσία και θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς και πότε σκοπεύετε να το συζητήσετε αυτό το θέμα. Λέτε ότι το έχετε θέσει ως στόχο. Ίσως λοιπόν κάποιο σύντομο σχόλιο και η ερώτηση πολλά συζητήθηκαν κατά πόσο θα πρέπει Όλα αυτά θα είναι ε, δωρεάν. Όχι, θα ήθελα την απάντησή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ που αναφέρετε αυτό το θέμα. Έγινε πολλή εργασία για αυτό το θέμα που αφορά τους καταναλωτές. Ε, το έθεσα λοιπόν ως μία τις τρεις προτεραιότητες της δραστηριότητάς μου για το 2012. Δεν πιστεύω στην αυτορύθμιση των αγορών. Στην... η ελευθέρωση έκανε πολλές ζημιές. Η απορρίθμιση σε ορισμένες ε, περιπτώσεις έκανα την επιλογή να προτιμήσω με τους συναδελφούς μου το συμβόλαιο και όχι τον περιορισμό. Αυτό συνέβη για του βασικού τραπεζικού λογαριασμού όπου ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να δράσουν. Θα το θυμάστε. Το ίδιο ίσχυσε και για τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών, κάνοντα έκκληση στην καλή θέληση των τραπεζών. Και στι δύο περιπτώσει αυτέ, εγώ εξέφρασα την απογοήτευσή μου είδα ότι η μέθοδος των συμβάσεων, των συμβολέων δεν ήταν επαρκής για τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχουμε σήμερα ένα μέρος των απαντήσεων. Θα κάνουμε την αξιολόγηση του συνόλου των απαντήσεων πριν το τέλος Ιουλίου και για να σας απαντήσω με ακρίβεια στην ερώτησή σας προτείνω μια νομοθεσία δεσμευτική διότι το συμβόλαιο δεν ήταν επαρκές πριν από το τέλος του έτους, ε, πριν το τέλος του 2012. Ε, πιθανότατα θα κάνουμε το ίδιο και για τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών και για την κινητικότητα των λογαριασμών που είναι απολύτως αδύνατη σήμερα ή εξαιρετικά δύσκολη για τους πολίτες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν τραπεζικούς λογαριασμού. Γι' αυτά λοιπόν τα τρία θέματα θα προχωρήσουμε σε πιο δεσμευτικά μέτρα. Right, thank you. Um, I Ευχαριστώ. Να κάνουμε τώρα ομάδες των τριών ερωτήσεων. Πρώτη ομάδα είναι Σόφι, Άρλιν Μακάρθι και Φιλίπ Λάμπερτς. Δεύτερη ομάδα, Άννη Ποδηματά, Σάντσες Προζέντο και η τέταρτη ομάδα Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο και τον ξέχασα. Πρώτη ομάδα με τη Σόφη. Ευχαριστώ. Άργησα να έρθω στην αίθουσα, κύριε Επίτροπε, αλλά ήμουν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία ξεπέρασε το ωράριό της, για τα βιοκαύσιμα και την ενέργεια. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πρωτοβουλίες σας όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και χαίρομαι που θα... είμαι στην ίδια ομάδα με τον Φιλίπ Λάμπερτς γιατί θεωρώ ότι όπως εργαστήκαμε μαζί και με πολύ υποδομικό τρόπο για τα θέματα των κοινωνικών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κεφαλαίου βρίσκω ότι η προληπτική, θα έλεγα, δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Μέχρι τώρα είχαμε μία πολιτική μάλλον που αντιδρούσε στα γεγονότα της αγοράς. Σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, έχει αντιστραφεί αυτή η τάση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα αρκετά νωρίς, με ένα πολύ φιλόδοξο κείμενο, το οποίο αντιμετωπίσαμε με πολύ θετικό τρόπο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτον, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και δεύτερον να δημιουργήσουμε μία αγορά ευρωπαϊκή στον τομέα των επενδύσεων ε, στον τομέα αυτό της αλληλεγγύης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Επίτροπε, ποια είναι η άποψή σας Όσον αφορά την ενσωμάτωση αυτής της προσέγγισης σε μια πολύ γενικότερη πολιτική για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας νέος τομέας ο οποίος θα δημιουργήσει πλούτο, ο οποίος θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει αυτόν τον τομέα στη γενικότερη πολιτική της πρέπει να δοθούν κίνητρα, φορολογικά κίνητρα κατά την άποψή μου, κίνητρα για περισσότερες επενδύσεις στον ε, κοινωνικό τομέα, ένα ευρωπαϊκό σήμα, ευρωπαϊκό λάμπελ και τρόπους πρόθεσης επικοινωνίας όσον αφορά αυτόν τον νέο τρόπο χρηματοδότησης της οικονομίας. Άλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο διατραπεζικό σύστημα και στα επιτόκια καθώς και τις διάφορες φήμες για στρέβλωση του ανταγωνισμού, χειραγώγηση και συμφωνίες. Οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει και στις οποίες εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχουν προχωρήσει. Θα ήθελα ενδεχομένως να ακούσω από εσάς πώς έχει αυτή η έρευνα. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια στις αγορές, δεν θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι χειραγωγήσεις και θα ήθελα να ξέρω όσον αφορά την οδηγία για την διαφάνεια και επειδή είμαι εισηγήτρια για την νομική επιτροπή, θα ήθελα να σας ζητήσω να προχωρήσετε. Μήπως όμως είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές εταιρείες που υιοθετούν σήμερα μέτρα βάσει του Transparency International. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τους τομείς όπως αυτών της εξορρυκτικής βιομηχανίας ή της ε, υλοτόμησης. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας πω ότι αναφέρατε μία πράσινη βίβλο για τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Εγώ θα ήθελα να σας πω, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε την οικονομία καζίνο. Δηλαδή, μιλήσατε για το trading υψηλής συχνότητας. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Αυτό που είναι κερδοσκοπία και οικονομία καζίνο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αφήνουμε από τη μία αυτού του είδους τις πρακτικές και από την άλλη να προσπαθούμε να ε, μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να σας πω. Αναφερθήκατε στο shadow banking. Πρόκειται για έναν τομέα τον οποίο θα πρέπει να επεξεργαστούμε με τα νέα μέτρα, με το σεμινάριό σας και με τις εργασίες που γίνονται στην Επιτροπή θα καταλήξετε σε κάποιο νομοθετικό κείμενο. Euh, Ευχαριστώ τη Σοφία Κονή για την ενθάρρυνσή της όσον αφορά αυτό τον μεγάλο τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας όπως λέγεται, που για την πραγματική μας οικονομία είναι το 15-16% καθώς και των θέσεων απασχόλησης. Μιλούμε λοιπόν για επικερδείς επιχειρήσεις δεν μιλούμε για ενώσεις ή για κοινωνικές υπηρεσίες. Μιλούμε για επιχειρήσεις που έχουν αλληλέγγυο και ηθικό χαρακτήρα, αν θέλετε, αν μπορώ να το πω έτσι, φύση, και προσωπικό το οποίο θέλει να φέρει σε πέρα αυτό το ηθικό έργο και επιτελεί έργο στις αγορές και κερδίζει ένα μέρος της αγοράς. Πρόκειται για διαφορετικές λοιπόν επιχειρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και αυτό είναι και ο στόχος αυτού του ταμείου. Πράγμα το οποίο ε, είναι μια ιδέα που μου έδωσαν αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Και βεβαίω δεν θα σταματήσουμε εδώ και συμμερίζομαι και την δική σα πρωτοβουλία. Αυτό εξάλλου με τον κύριο Αντόρ και με τον κύριο Ταγιάννη ε, ως θέμα το προωθήσαμε στα πλαίσια μίας ε, διάσκεψης που έγινε και με την παρουσία του καθηγητή Ονούς με την, το Νοέμβριο τον προηγούμενο με την παρουσία 1.200 συμμεταχόντων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την κατάλληλη πλαισίωση και την κατάλληλη νομική ε, βάση για να συνοδεύσουμε αυτού το είδους τις εταιρείε. Γι' αυτό εμείς κάνουμε προτάσεις όπως φερρυπίν αυτή που κάναμε για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ορατότητα στον τομέα αυτό. Και αυτό θα επιτευχθεί και μέσω αυτών των σημάτων των ευρωπαϊκών, των διαβατηρίων. Βλέπω με μεγάλη προσοχή τι γίνεται γύρω μου σε πολλές χώρες, κυρίως και στην χώρα σας κυρία Πρόεδρε, όπου και οι συντηρητικοί και οι εργατικοί πήρανε τις κατάλληλες αποφάσεις για το social business. Και πολλές φορές γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν κάποια κεφάλαια τα οποία κοιμούνται στις τράπεζες για να βοηθηθεί ο κόσμος. Όλες αυτές οι ιδέες είναι ενδιαφέρουσες λοιπόν και θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε στην νομική πλαισίωση στην ε, χρηματοπιστωτική διευκόλυνση και στην ορατότητα όλων αυτού του εγχειρήματος. Σας... Όσον αφορά τώρα τα μπόνους και τα άλλα θέματα που ε, αναφέρατε, ε, συμφωνώ, δεν μπορώ για τις έρευνες αντιθέτως να πω πάρα πολλά θέματα αντικειμενικά σχόλια δημοσίω που μπορώ να κάνω για έρευνε οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Και από νομικής πλευράς θα δω εγώ ποια είναι τα περιθώρια που έχουμε για να μπορέσουμε να σα δώσουμε κάποια άλλη φορά ε, σε εσά και στην προεδρό σα κάποιε πληροφορίε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω για αυτέ τι τρέχουσε έρευνε που διεξάγονται κανένα σχόλιο. Φιλίπ Λομπέρ. Αναφέρθηκατε στο country per country. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Πήρε την πρωτοβουλία να πάει αρκετά μακριά η Κομισιό. Μακρύτερα από ό,τι περισμένανε κάποιοι. Διότι προτείναμε διαφάνεια για 600 εταιρείε εισηγμένε ή όχι τη εξορρυκτική βιομηχανία και τη βιομηχανία στον τομέα τη ηρετομία. Προχωρούμε σταδιακά. Και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε αυτό τον τομέα του πεδίου εφαρμογής. Τώρα μπορούμε να πάμε πιο μακριά, να προχωρήσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλώς προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που είχαν υποβάλει κυβερνήσεις, κυρίως αφρικανικών κρατών και διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αυτοί οι οποίοι είχαν κυρίως υποφέρει από αυτή την έλλειψη διαφάνειας στην εξορρεκτική βιομηχανία. Και το ίδιο έγινε και στον τομέα της υλοτομίας. Ας αρχίσαμε από αυτούς τους τομείς. Ας προχωρήσουμε. Δεν είναι όλα κερδισμένα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να επιβάλλουμε για κάθε σχέδιο χωριά, για κάθε χώρα χωριστά την διαφάνεια στους δύο αυτούς τομείς και θα προχωρήσουμε μετά. Αναφέρεις το καζίνο, Φιλίπ. Και εγώ, κύριε Λαμπερ, είπα προηγουμένως και το έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η εμπιστοσύνη την οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσει να ξαναρχίσει να λειτουργεί πραγματική η οικονομία βασίζεται σε σταθερές και διαφανείς βάσεις. Δεν έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε αρχίσει όμως. Και χάρη στη δική σας εργασία και στην εργασία του Συμβουλίου, επίσης θα βελτιωθεί η κατάσταση του μεθόλου Τώρα, για το IFS Trading. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, ότι όντως δεν πάει πολύ μακριά και πολύ γρήγορα η Κομισιόν στο θέμα αυτό. Το δέχομαι. Προσπαθώ όμως να κάνω τα πράγματα με τρόπο έξυπνο και όντας και ρεαλιστής, για να προχωρήσουμε. Όχι για να μπλοκαριστούμε κάπου. Το θέμα αυτό μπορούμε μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι και για το, για λογαριασμό μας να το χειριστούμε χωρίς να ασχοληθούμε με το τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Εγώ συνεργάζομαι αυτό το θέμα με την κυρία Σαπύρο και τον πρόεδρο του FCF που επίσης, επίσης τους απασχολεί το θέμα αυτό. Και ο κύριος και η κυρία Σαπύρο ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το trading υψηλής συχνότητας. Και προσπαθώ να δω τι μπορούμε να αποκομίσουμε συνεργαζόμενοι και με τους Αμερικανούς στον τομέα αυτό. Θα θέσουμε σε εφαρμογή όλα αυτά τα μέτρα που είναι αρκετά επαχθή αν κρίνω από την αντίδραση ορισμένων κυρίως από αυτούς που επιδίδονται σε αυτή τη δραστηριότητα και από αυτούς οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο και μαζικά δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι. Στο ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε πέρα της εργασίας ανάλυσης πραγματογνωσύνης για το shadow banking και όσον αφορά την δομική διαχείριση στις τράπεζες. Για τον διαχωρισμό των κινδύνων και για το trading high frequency προσπαθούμε κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού για αυτά τα θέματα. Θέλω να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα, ανάλογα με, την, το καθένα και την ε, βαρύτητά του και να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε, ανάλογα με το τι ρίσκο σημαίνει και αυτό για το κάθε θέμα. Θα κάνουμε λοιπόν κάτι και καταλήξουμε και στην νομοθεσία, φαντάζομαι, με το shadow banking. Okay. We're just waiting for Ωραία. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διερμηνία. Παύλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με ευχαρίστηση άκουσα τις περισσότερες παρατηρήσεις σας και σας παρακαλώ συνεχίστε να εργάζεστε προς αυτή την κατεύθυνση που είναι σωστή. Εσείς ε, Είπατε ότι θέλουμε πραγματικά όλε τι χρηματοπιστωτικέ δραστηριότητε να στα πλαίσια πραγματική οικονομία. Συμφωνώ μαζί σα. Επίση, στα πλαίσια κάποιων εβδομάδων είπατε ότι θα υπάρξει έλεγχο στα τραπεζικά συστήματα, τα shadows, τα περίφημα. Σα ε, ε, υποστηρίζουμε επίση σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πιστεύω ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση του πραγματικού τραπεζικού συστήματος, διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπε η κυρία Φεραίρα, χρειάζεται ρευστό στις αγορές για να κινηθούν οι οικονομίες. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ανάκτηση της οικονομίας και αηφόρο ανάπτυξη. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν της ε, αναδιάρθρωσης ε, της οικονομίας, πιστεύω ότι πολλά πράγματα γίνονται ατακτά. Ε, ασυντόνιστα, αν θέλετε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Παρά το γεγονό ότι δεν είναι τη δική σα ε, αρμοδιότητα, ξέρουμε ότι γίνανε stress test για τι τράπεζε, ξέρουμε ότι ίσω δεν γίνουν άλλα τέτοια είδου τεστ. έχουμε όμω την εντύπωση, και συγγνώμη που το λέω, ότι τα πράγματα έχουν γίνει με ανοργάνωτο τρόπο. Θα σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Επίτροπε, πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα πραγματικά χρηματοπιστωτικό σύστημα αναδιαρθρωμένο στο οποίο θα ρέει το χρήμα για να μπορέσει να υπάρξει αηφόρος ε, ανάπτυξη της οικονομίας και αναδιάρθρωση της οικονομίας. Ευχαριστώ. Γιάννη. Thank you, Sharon. Ευχαριστώ, Σάρων. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για τις παρατηρήσεις σας. Ε, εδώ είμαι. Ευχαριστώ επίσης ε, που επιβεβαιώνετε για άλλη μία φορά τη δέσμευσή σας η οποία είναι και η δική μας δέσμευση, η δημιουργία υγιών και σταθερών βάσεων για την αδρομολόγηση, την επαναδρομολόγηση θα έλεγα του χρηματοπιστωτικού τομέα ε, στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη δική μου ερμηνεία, κύριε Επίτροπε, αυτό σημαίνει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο υπογραμμίστηκε από πολλούς συναδέλφους. Είναι επίγον το ζήτημα, ειδικότερα υπό τις τρέχουσες συνθήκες, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες και γρήγορες λύσεις. Το σημείο αυτό υπογραμμίστηκε από τον συνάδελφο Φιλίπ Λαμπέρτ στην Ελίζα Φεραίρο επίσης. Η πράσινη βίβλος που αναγγείλατε φοβόμαστε, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να παράσχει γρήγορε και συγκεκριμένες λύσει. Η ερώτησή μου είναι η εξή: Εν αναμονή αυτή της πρωτοβουλία για την πράσινη βίβλο υπάρχουν μήπω άλλα μέσα, άλλε προτάσεις, άλλε πρωτοβουλίε που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα ώστε να εξασφαλίσουν για παράδειγμα ότι η ρευστότητα που, του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία, ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος της κρίσης και σας διαβεβαιώ ότι για παράδειγμα σε εμά στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οδηγούνται σε μια διαδρομή τρόμου προς την χρεοκοπία λόγω των προβλημάτων έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Και εν συντομία το δεύτερο σημείο ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για την υιοθέτηση μια, ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις ε, στο ΕΚΟΦΗΝ, στο Κοινοβούλιο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε ακούσει κάποια επιχειρήματα από όσου είναι αντίθετοι σε αυτό το φόρο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένας φόρος ο οποίος θα υλοποιούνταν ε, είτε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ακόμη χειρότερα σε επίπεδο ευρωζώνης θα μπορούσε να δημιουργήσει μειονεκτήματα σημαντικά για το χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη και πιο συγκεκριμένα συμφωνείτε με όσους λένε ότι αυτός ο φορός θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα, τα αποταμιευτικά, στις αποταμιεύσεις. Ευχαριστώ. Αντολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, όταν σας άκουσα, είχα την εντύπωση ότι η δική σας ε, ότι αυτή η θητεία είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη, διότι υπάρχουν εξαιρετικέ πρωτοβουλίε, οποίε μιλήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να σα συγχαρώ, διότι συνεργαζόμαστε και είμαστε πάρα ε, πολύ ε, ευτυχεί γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα ενηθυπόθηκα δάνεια, πρέπει να μιλήσουμε για υπεύθυνο δανεισμό. Και στην παρούσα κρίση θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα. Με ικανοποιούν οι προτάσεις οι οποίες έγιναν στις συζητήσεις που γίνεται για τα ενυπόθηκα δάνεια, που είναι αυτό του διαχωρισμού του ρίσκου. Πιστεύω ότι άρχισε μια διαδικασία η Κομισιόν σε αναφορά τα προβλήματα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τα προβλήματα των καταναλωτών που έχουν οικονομικά προβλήματα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, τι κάνετε σε αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση και να μας πείτε τι κάνετε επίσης και με τα ιδρύματα ή με τους οργανισμούς που είναι υπερχρεωμένοι αυτή τη στιγμή. Πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό εσείς στην υπηρεσία σας. Ε, ο κύριο Άλμπα, όπως και η κυρία Ποδηματά προηγουμένως, ανέφερε την πραγματική οικονομία, ειλικρινά. Χαίρομαι, διότι μετά από όλη την δουλειά που έγινε εγκαρσίως για την ρύθμιση των διαφόρων τομέων ε, προληπτικά, θα πρέπει να ασχοληθούμε τώρα με την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Χαίρομαι λοιπόν που το αναφέρετε εσείς και δεν εκπλήσωμα. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει την ρυθμιστική δουλειά που έχουμε αρχίσει να την ολοκληρώσουμε, διότι δεν έχουμε τελειώσει και θα πρέπει πολλές φορές να καταλάβουμε τι γίνεται και σε κάποιους άγνωστους για μας τομείς. Το shadow banking φερρυπίν, που πραγματικά αναπτύχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι υπεύθυνο το 30-35% των συναλλαγών. Τώρα, πριν από κάτι για το shadow banking. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν ενοχοποιώ το τομέα. Πιστεύω ότι πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον μη ρυθισμένο ή κακά ρυθισμένο τομέα κάνουν χρήσιμα πράγματα για την οικονομία. Και πολλές φορές προσφέρουν τη χρηματοδότηση την οποία για χ ή δεν μπορεί να παράσχει το τραπεζικό σύστημα. Δεν αναχοποιώ λοιπόν κανέναν ή δεν κάνω κρίσεις επί των θεμάτων. Απλώς θέλουμε να υπάρχει εποπτεία του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο τομέας και να υπάρχει διαφάνεια. Αναφέρατε τα stress test, τα οποία γίνονται όπως λύσαμε υπό την ηγεσία των τραπεζών στην Ευρώπη. Θα μπορούσε στο μέλλον να υπάρχουν και άλλα, παρά το γεγονό ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο άμεσα, αλλά η Ευρωπαϊκή Αρχή των Τραπεζών είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για το πότε και το πώς. Κάτι σημαντικό μου ρωτήσετε. Πότε θα μπει τάξη στον τραπεζικό ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την δουλειά την οποία επιτελούμε. Αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, γύρω στα 15 κείμενα τα οποία βρίσκονται τώρα στην ε, ε, νομοθετική ε, οδό, αν θέλετε. Όταν θα ψηφιστούν, θα είμαστε λίγο πιο βέβαιοι ότι μπορούμε εσωτερικά ή εξωτερικά να εποπτεύουμε καλύτερα, να ελέγχουμε καλύτερα ότι υπάρχουν καλοί κανονισμοί, καλές ρυθμίσεις, διαφάνειες κτλ. Δεν έχουμε φτάσει όμως σε αυτό το στάδιο ακόμη. Ας δουλέψουμε σωστά και ας μην ξεχνάμε και κάποια πράγματα. Κυρία Ποδηματά, είπατε προηγουμένως ότι ορισμένοι φοβούνται ότι ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν υπάρχει ακόμη αυτός ο φόρος, αλλά αυτό που δημιούργησε πρόβλημα είναι η χρηματοπιστωτική κρίση και ο ανεύθυνος τρόπος με τον οποίο ενήργησαν κάποιες τράπεζες. Κάποιες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες. Ξέρουμε πώς ενήργησαν. Και βεβαίως ήξερα ότι δεν πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και να εφαρμόζονται κάποιοι κανόνες ηθικής, ώστε οι εταιρείε που περιμένουν και οι καταναλωτέ και οι πελάτες που πρέπει να περιμένουν κάτι από τι τράπεζε, να το περιμένουμε εμπιστοσύνη από τις τράπεζές τους. Δεν έχουμε φτάσει λοιπόν στο τέλος των προσπαθειών μας και ας μην ξεχνούμε κάποια πράγματα παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα νομοθετήσουμε και ποια θα είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος της νομοθεσίας που θα κάνουμε κατά τη κρίσης. Τώρα, η πράσινη βίβλος είναι ένα μέσο να γίνει δημόσια διάλογος και διαφούλευση. Εμείς ε, δεν δεν είμαστε παντογνώστες, Πρέπει να δούμε όλοι από κοινού πώς θα μελετήσουμε το θέμα των ε, υποδομών, της χρηματοδότησης των έργων υποδομής, της οικολογικής διάστασης η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί στην ε, ανάπτυξη οικονομίας, ώστε να είναι καλύτερα οι επόμενες γενιές. Αυτό βλέπω εγώ όταν μιλούμε για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση οικονομίας. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι τα νομοθετικά μας έργα θα πρέπει ίσως να είναι πιο άμεσα. Εγώ το είπα και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα στοχεύουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης. Τα project bonds μπορούν να δημιουργηθούν σε μερικούς μήνες. Εάν υπάρχει μεταξύ των Ευρωπαίων κλίμα εμπιστοσύνης, δεν χρειαζόμαστε τρία-τέσσερα χρόνια για να μπορέσει να υπάρξει ένα μέσον δανεισμού ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις έργα υποδομής στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις ψηφιακές τεχνολογίες κτλ. Όσον αφορά τη ρευστότητα, τα μέτρα που αφορούν τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνουμε και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα να βοηθήσει μέσω διατραπεζικού δανεισμού τις άλλες τράπεζες για να αρχίσει να κινείται η οικονομία. Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία διέθεσε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην Ευρώπη σε 800 τράπεζες περίπου. Πάρα πολλές κυβερνήσεις υποστηρίζουν την ιδέα αυτή του φόρου των ε, ε, ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν έχουν όμως οι πάντες συμφωνήσει. Ο κύριος Εμέτα ασχολείται με αυτό το θέμα και πρότεινε δύο ποσοστά πολύ χαμηλά, πράγμα που για μένα είναι κάτι το οποίο από ε, πλευράς οικονομιών μπορεί να αποφέρει 57 εκατομμύρια ευρώ, δις ευρώ, ε, πολιτικά είναι σωστή και μπορεί να βοηθήσει τους πάντες. Δεν μιλώ μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλους τους Ευρωπαίους πρέπει να δώσουμε σε όλους ε, το μήνυμα ότι αυτό το οποίο ζητούμε είναι δίκαιο, είναι σωστό και πρέπει κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, τα μπόνους των τραπεζών, τα πολύ υψηλά και τα δικαιολόγητα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εμείς να τα επιτρέψουμε. Και είναι δίκαιο αυτό το θέμα του φόρου. Και θα μπορέσουν έτσι να κάνουν μια προσπάθεια οι πάντες για να μην επανέλθουμε με μεγάλες ζημίες σε μια φάση προστατευτισμού. Ο κύριος Βασέντο ανέφερε τα ενυπόθηκα δάνεια, αλλά πιο γενικά το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Για το θέμα των, ε, της υπερχρέωσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Με τον κύριο Ταγιάννη θα μιλήσω για το θέμα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα όσον αφορά τους καταναλωτές. Ό,τι κάνουμε με τα PRIPS, με, τις με τα εγγυημένα δάνεια, το κάνουμε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την υπερχρέωση των πολιτών, για να αμβλύνουμε το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να είναι σωστά ενημερωμένοι οι πολίτες για τους κινδύνους που υπάρχουν, για τα προϊόντα, τα τραπεζικά τα οποία, στα οποία θα προσφύγουν και στην προστασία που θα τους προσφέρουμε τελικά. Αυτή είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας για το 2012. Επόμενος ομιλητής, Πασκάλ. Θα χρησιμοποιήσω και του ούντο το χρόνο ομιλίας, εντάξει. Α, δεν μπορώ, δυστυχώς. Κύριε Μπαρνιέ, σας χαιρετώ. Καταρχήν έχω δύο ερωτήσεις. Είχατε δεσμευθεί πριν από λίγο καιρό εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, όσον αφορά τα CDS. Ξέρετε ότι όσον αφορά τις ε, συναλλαγές αυτές έχουμε θέσει κάποιους ε, περιορισμούς και κάποιους κανονισμούς για τα CDS, αλλά όχι όσον αφορά την ε, πώλησή τους. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι αν υπάρξει ένα επεισόδιο και ενεργοποιηθούν αυτά τα CDS, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Ξέρετε ότι η λύση θα μπορούσε να είναι να γίνουν κάποια stress test όσον αφορά τους εκδότες CDS, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μπορούν σε περίπτωση που ενεργοποιούνται τα CDS να πληρώσουν. Είδαμε, παραδείγματος χάρη με την EAG και την κρίση των subprimes, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν σε θέση η EAG να επιστρέψει τα ποσά από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκαν τα CDS. Μία άλλη ερώτηση. Διάβασα στην Financial Times ότι υπήρξε μία συναλλαγή μεταξύ της ε, δικής σας ε, θέσης μεταξύ κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ερωτώ λοιπόν, σας στηρίζει 100% ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Νίκολας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας αισθανθήκατε την ανάγκη να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα συναδέλφων που θεωρούσατε ότι εκκρεμούσαν πλήρεις απαντήσεις μου δίνετε λοιπόν την αφορμή να σας ξαναθέσω ένα ερώτημα που σας το έχω θέσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια και απάντηση δεν έχω πάρει. Και αυτή η επιμονή έχει να κάνει, διότι το πρόβλημα αυτό συνδέεται με τα ασφαλιστικά ταμεία, με την αξιοπιστία σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα, αλλά λυπάμαι και με τη δική σας προσωπική αξιοπιστία και την αξιοπιστία της Κομισιόν. Είναι το πρόβλημα της παράνομης πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, στην Deutsche Telekom. Δεν έκανε δημόσια δημοπρασία, με συνέπεια να πληγούν ασφαλιστικά ταμεία και μικρομέτοχοι. Σας κάνω ερωτήσεις δυόμιση χρόνια. Λέτε ότι διαπιστώθηκε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και πέραν τούτου τίποτα. Η συνέχεια ο κύριος Βενζέλος ως αντιπολίτευση είχε καταγγείλει αυτή τη συμφωνία, ως υπουργό στη Βουλή λέει ότι ήταν παράνομη αυτή η συμφωνία, αλλά στη συνέχεια πώλησε ένα μεγάλο μέρος των μετοχών, το υπόλοιπο, στην Deutsche Telekom. Συνεχίστηκε δηλαδή αυτό. Σας ερωτώ λοιπόν, ήταν παράνομη αυτή η πώληση. Δεύτερο, αν ήταν παράνομη εσείς και το διαπιστώσατε παραβίαση της, ε, ε του 25-2004. Τι κάνετε να την ακυρώσετε. Τρίτη ερώτηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ποιον εξυπηρετείτε, ποιον υπερασπίζεστε. Την Deutsche Telekom που κέρδισε εκατομμύρια σε βάρος των μικρομετόχων, σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Δώστε μου σας παρακαλώ μια απάντηση και σας ξαναλέω είναι θέμα και προσωπικής σας ευθύνης, ευθύνης της Κομισιόν και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Αστρίντ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν ήθελα αρχικά να μιλήσω όσον αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διότι δεν αποτελεί δικό σας φάκελο, είναι φάκελο του συναδέλφου σας. Αλλά φυσικά, καθώς η Επιτροπή λειτουργεί συλλογικά, έχετε κι εσείς φυσικά το μερίδιο, το δικό σας μερίδιο ευθύνης ε, όσον αφορά την πρόταση που μας υπευλήθη για την εισαγωγή αυτού του φόρου όπως είπε η συγγήτρια κυρία Ποδηματά ε, και έκανε αυτή την ερώτηση ήθελα και εγώ να μάθω εάν αυτά που διάβασα στον τύπο μετά από το τελευταίο Συμβουλίο Υπουργών σε σχέση με αυτό το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από όσο κατάλαβα υπό τη μορφή υπό την οποία την έχετε προτείνει έχει πεθάνει γιατί εμένα μου έκανε έκπληξη που άκουσα από μέρους σας ότι δεν βλέπετε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την, ε, από την μετατόπιση εγώ πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στον ε, σοσιαλιστικό τύπο του Λουξεμβούργου Δυστυχώ δεν το έχω μπροστά μου και δεν μπορώ να πάω να το ψάξω να το βρω στο γραφείο που δείχνει τις δυσμενείς επιπτώσεις ειδικότερα σε θέματα μετεγκατάστασης ε, που θα απέραν από την πρόταση της ε, ε, Κομισιόν λόγω του φαινομένου χενοστιβάδας που επιφέρει αυτός ο φόρος. Θα ήταν ε, μοιραίο για μεγάλο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι εξάλλου θα σας στείλω και αυτό το άρθρο. Ευτυχώς ο δικός μας υπουργό Οικονομικών επίσης ε, κατάλαβε παρότι ο Πρωθυπουργό μας εξακολουθεί να λέει άλλα είχε πει τουλάχιστον εκείνη την εποχή άλλα πράγματα έπαιρνε αυτού διότι ακούσαμε από την Κομισιόν ε, ε, να λέει ότι ο δικός μας ο Πρωθυπουργός είναι υπέρ του φόρου, ωστόσο ο Υπουργός Οικονομικών μας τώρα, οικονομικών μας τώρα του έδωσε να καταλάβει ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις, ε, κυρίως μάλιστα και για τον προϋπολογισμό του Λουξεμβούργου από μια τέτοια υπόθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να δούμε με τρόπο κάπως πιο αντικειμενικό, να δείτε και εσείς κάπως πιο αντικειμενικά τις πιθανές επιπτώσεις της δικής σας πρότασης. Ε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε ένα τέτοιο, φόρμο, ε, ένα τέτοιο φόρο, αλλά η δική σας πρόταση φαίνεται να μην μπορεί να έχει εφαρμογή. Ε, επίσης, ε, φαίνεται να έχει επιπτώσεις απαράδεκτες. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν ε, καλό θα ήταν ε, να αποσύρει αυτή την πρόταση και να μελετήσει εναλλακτικέ προτάσει, τι οποίε θα μπορούσε να κάνει για την εισαγωγή ενό φόρου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η οι περισσότερες πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι η καλύτερη λύση θα ήταν παγκόσμιος φόρος. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο είναι ουτοπικό, αλλά αν θέλουμε φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να εφαρμόσετε τους 27 χωρίς εξαιρέσεις επειδή κάθε κράτος μέλος φυσικά είναι ελεύθερο να δημιουργήσει ένα τέτοιο φόρο. Δεν πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να πιστεύει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να τους δώσει άδεια. Εάν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε θέλουν να δημιουργήσουν ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στη Γερμανία, έχουν το ελεύθερο να το πράξουν αύριο. Και προχθές ήταν ελεύθεροι να το πράξουν. Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης έχει την ελευθερία να το πράξει. Δεν πρέπει λοιπόν ε, να νομίζουμε ότι οι χώρες ε, που θέλουν να υιοθετήσουν ένα τέτοιο φόρο χρειάζονται την Ευρώπη. Μπορούν κάλλιστα ε, να το πράξουν μόνος τους. Είναι αυτόνομες, έχουν την αυτοκυριαρχία τους και μπορούν να το πράξουν. Ε, αν πιστεύουν ότι τη συμφέρει, εμένα δεν με πειράζει να το πράξουν, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι χώρες που θα υποστούν τεράστιες επιπτώσεις για την απασχόληση και τη ε, δημόσια έσοδα θα πρέπει επίσης να έχουν την ελευθερία να μην υιοθετήσουν ένα τέτοιο φόρο. Θα ήθελα να σταματήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι θέμα του κατά ποιος, ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά. Όποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Ο κύριος Γιούνκερ όμως πρώτος ε, είχε κάνει την πρόταση να υιοθετηθεί στην Ευρωζώνη. Δεν ήταν η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Σόιμπλε πρώτος ο κύριος Γιούνκερ. Μήπως να μιλήσετε πρώτα με τον κύριο Γιούνκερ στο Λουξεμβούργο. Ίσως αυτό θα είναι πιο εύκολο από ότι εδώ. Μπορώ να απαντήσω, συγγνώμη, μία πρόταση. Πριν από ένα χρόνο και παραπάνω είχε κάνει εκείνη την ομιλία του υπέρ της εισαγωγής αυτού του φορού επειδή ο Υπουργός Οικονομικών του του έλεγε ε, και τότε ήταν αντίθετος. Πιστεύω κύριε Γκίγολτ, είναι πολύ εύκολο και εγώ θα μπορούσα να είμαι υπέρ. Γιατί ξέρω δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν είμαι τόσο υποκρίτρια. Okay. Uh, λοιπόν, να απαντήσει ο Επίτροπος. Βεβαίως δεν είναι όλα τα θέματα... Ε, αρμοδιότητά του, αλλά όντω μπορεί οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί να αλλάξουν άποψη για κάποια θέματα. Συμβαίνει αυτό. Ναι, αλλά όπως είπε η κυρία Λούλινγκ, με πάθος, είμαστε συλλογικό όργανο, δεν είμαστε, αν θέλετε, ένας συμπαγής οργανισμός. Γι' αυτό και εγώ είμαι αλληλέγγυος με αυτή την πρόταση ο συντονισμός και η αναρμόνιση σε κάποιους τομείς της φορολογίας είναι ο σκοπός μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με 27 διαφορετικές ε, φορολογικές βάσεις όσον αφορά ε, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και όπως ξέρετε θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, η μόλυνση να έχει σαν αποτέλεσμα πολύ αυστηρότερες ε, κυρώσεις, έτσι ώστε να σταματήσει. Έχετε δίκιο πάντως ότι το θέμα της φορολόγησης των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι κάτι το δίκαιο και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι και να κατανείμουμε ισομερός τις προσπάθειες. Σήμερα οι λαοί της Ευρώπης κινδυνεύουν να αντιδράσουν, να εξεγερθούν και θα έχουμε ε, την εκμετάλλευση αυτής της αντίδρασης από δημαγωγικές ε, και εξτρεμιστικές ε, ε, πολιτικές δυνάμεις. Έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να επιβληθεί παγκοσμίως ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας τέτοιος φόρος. Όπως ξέρετε, για κάποιες ε, συναλλαγές υπάρχουν ήδη τέλη και φόροι. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, έχει επιβάλει κάποιο φόρο στι συναλλαγέ χωρί να ζητήσει την άδεια από κανέναν. Το ίδιο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι λοιπόν ε, θέμα απαγορευμένο, αλλά όντω πρέπει να επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είναι πιο δίκαιο αυτό ο φόρο. Μιλήσατε για την ρύθμιση των ε, πωλήσεων των ε, CDS. Αυτό το κάναμε χάρη σε εσά εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την αγορά αυτών των ε, προϊόντων, των CDS. Η διαχείριση του κινδύνου για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βεβαίως είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα και η επίλυση των τραπεζικών κρίσεων. Κύριε Κομφά, θα σας απαντήσω. Οι εκδότες CDS είναι σε μεγάλο βαθμό τράπεζες. Τράπεζες που θα υποβληθούν στις απαιτήσει και στους κανονισμούς όσον αφορά το κεφάλαιο και ζήτησα από την ΕΣΜΑ να επεξεργαστεί το θέμα αυτό, λαμβάνοντας την ελληνική εμπειρία υπόψη της και θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και είτε να γίνουν stress test, είτε για τους εκδότες ιδιές που δεν είναι τράπεζες, να ελέγξουμε όσον αφορά την αντοχή τους με κάποιον άλλο τρόπο. Μία άλλη ερώτηση. Ναι, Είπατε ότι εσείς διαβάζετε το Financial Times. Η κυρία Λούλινγκ διαβάζει σοσιαλιστικές εφημερίδες από το Λουξεμβούργο. Και εγώ διαβάζω το σοσιαλιστικό τύπο, διαβάζω και το Financial Times. Όχι όμως ε, τυφλά, διότι πολλές φορές δεν είναι και σωστές οι πληροφορίες. Εγώ σας το λέω πολύ απλά. Πρώτη φορά ακούω αυτήν την ιδέα. Τι να σας πω. Προσπαθώ να ερμηνεύσω την παρατήρησή σας κύριε Κομφά. Θέλετε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, έτσι. Αυτό μου λέτε. Θα συνεχίσουμε. Βεβαίως, ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η εξωτερική πολιτική και ο τομέας της άμυνας. Τελειώνω με την τελευταία και αρκετά δύσκολη ερώτησή σας. Ξέρω ότι η ερώτηση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μου τίθεται κύριε Χουντή. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Βεβαίως δεν μπορώ να δικαιολογήσω τα πάντα, αλλά όντως ελήφθησαν κάποιες εξαιρετικές αποφάσεις για εξαιρετικές καταστάσεις. Μου λέτε να παρακολουθήσουμε την σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ιδιαίτερα λέτε ότι πρέπει να γίνει αυτό σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και θα γίνει ένας έλεγχος, μια αντικειμενική εξέταση. Η χώρα σας έχει υποβληθεί, έχει περάσει από πολλές δυσκολίες, σας έχουν επιβληθεί διάφορες ε, δύσκολες, ε, αν θέλετε, απαιτήσει από μέρους μας, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες παρανομίες. Ναι, σύντομα. Θέλω να θυμίσω στον Επίτροπο ότι η παρανομία για την οποία μιλάμε είναι πριν από την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα μου. Έγινε το 2008. Δεν δικαιολογείται στο όνομα της ειδική κατάστασης όλο το υπόλοιπο. Σας παρακαλώ πολύ. Τότε έγινε η παρανομία για την οποία συζητάμε και περιμένουμε απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά έλαβαν χώρα το 2008, παρότι η κρίση ξεκίνησε τότε. Η γρήγορη ιδιωτικοποίηση που λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα είναι κομμάτι της λύσης για μείωση της ε, κρατικής χρέωσης. Απλά αυτό που σας λέω είναι ότι οι δεδομένες καταστάσεις στη χώρα σας προσέχουμε, η και η δε, μέσω συγκεκριμένων μέτρων να μην προσθέσουμε δυσκολίες στις ήδη υπάρχουσες. Κάτι τέτοιο δεν θα δικαιολογούσε και ίσως εξηγεί κάποιες καθυστερήσεις, δεν ε, δικαιολογεί το να μην διαφωτίσουμε τις συνθήκες αυτής της ιδιωτικοποίησης. Εξακολουθούμε να μελετάμε αυτό το θέμα όπως το επιθυμείτε κύριε Χουντή και αυτό που σας είπα είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτών των μελετών που διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλατε εάν διαπιστωθούν παράνομες πρακτικές σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο θα εφαρμόσουμε τους κανόνες εγώ θα τους εφαρμόσω χωρίς ε, να, να κάνω χάρες ε, για διαδικασίες επί παραβάση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτρόπε. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας πιστεύουμε. Θα σας ξαναδούμε το φθινόπωρο, με βέβαια. Ευχαριστούμε. I think that uh, we will now have a short break for about minutes. Κάνουμε τώρα ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, διότι ο για το επόμενο θέμα δεν βρίσκεται ακόμη εδώ.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

Okay, we can resume. If we are... Okay, is, is everybody back, back in their seats? Right, we're now moving on to uh, agenda point 14. Το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης, που είναι ουσιαστικά γνωμοδότηση 20 κύριοι λόγοι ανησυχίας. Ο Έντουαρτ θα παρουσιάσει το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα καινούργιο θέμα με την έννοια ότι παρουσιάζουμε εδώ τις ανησυχίες άμεσα των Ευρωπαίων πολιτών και βάσει αυτού παρουσιάζουμε εδώ κάποιες ιδέες για το έγγραφο εργασίας της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται, αν θέλετε, για την ενιαία αγορά υπό το πρίσμα των πολιτών. Και εδώ παρουσιάζουμε τις δύο πιο κοινέ και συνηθισμένες ανησυχίες που έχουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Κάναμε λοιπόν μια ανάλυση όλες οι διαμαρτυρίες, όλες οι ανησυχίες των πολιτών και βασιστήκαμε σε υπηρεσίες για την απασχόληση, κέντρα ευρωπαϊκά και δίκτυα και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε όλες τις δυσκολίες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όταν θέλουν να εποφεληθούν από την ενιαία αγορά. Είναι, αν θέλετε, η εμπειρία των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Και βέβαια βασιζόμαστε επίσης και στο ευρωμαρόμετρο και σε άλλες μελέτες. Υπάρχουν δύο μεγάλες, ε, ε, αν θέλετε, ομάδες ε, διαμαρτυριών και ανησυχιών που προκύπτουν από μελέτες και από συζητήσεις. Είναι μια απεικόνηση, μια φωτογραφία της ενιαίας αγοράς με την εμπειρία των πολιτών επιτόπου, στην πράξη. Σε γενικές γραμμές λοιπόν επιβεβαιώνει εδώ ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών και της πραγματικότητας. Και αυτό προκύπτει από τρία χάσματα. Πρώτον, δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση. Ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά τους. Δεύτερον, υπάρχει ένα χάσμα όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή, λανθασμένη ή ελλειπής εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον, υπάρχει και ένα νομοθετικό χάσμα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά νομικά εργαλεία έτσι ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών από την ε, ενιαία αγορά και αυτών που μπορούν στην πράξη να αποκομίσουν και πώς μπορούν να επωφεληθούν. Η ΙΜΚΟ είναι η επί της ουσίας επιτροπή, η Ρετζίνα Μπάστος είναι η συγγήτρια. Εμείς απλώς ε, υποβάλλουμε μια γνωμοδότηση όχι επί των 20 ανησυχιών, αλλά μόνο επί αυτών που είναι περισσότερο αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, όπως παραδείγματο χάρη θέματα φορολογίας, ΦΠΑ, τραπεζικές υπηρεσίες, ε, συντάξεις, θέματα κληρονομιάς, φόρου κληρονομιάς και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όλα αυτά για άτομα στην Ευρώπη που θέλουν περισσότερη κινητικότητα, συναλλαγές διασυνοριακές, και κάθε άλλου είδους τέτοιες ανησυχίες ε, για εργοδότες και εργαζόμενους σε διασυνοριακό επίπεδο και επιχειρήσεις. Μεταξύ των σημείων που έχουμε επεξεργαστεί στη γνωμοδότησή μας είναι διαδικασίες για άνοιγμα λογαριασμού απλές, φιλικές προς τον ε, πολίτη, διπλή φορολόγηση και σε σχέση με του συνταξιούχους αλλά και σε σχέση με τη μεταφορά κεφαλαίων και την, το φόρο κληρονομιάς. Εδώ η Επιτροπή έχει υποβάλει απλώς μια σύσταση για τον φόρο κληρονομιάς και εδώ πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Επίσης το θέμα της γραφειοκρατίας αναφέρεται πολλές φορές. Καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξάρτητη συμβουλή σε σχέση με την χρηματοδότηση, ένας καλύτερος σχεδιασμός του καθεστώτος που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθούν παραδείγματος χάρη προβλήματα επιχειρηματικού κεφαλαίου, έλλειψη χρηματοδότησης και κεφαλαίων. Το θέμα του ΦΠΑ, της επιστροφής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις που έχουν ε, μια δραστηριότητα στο εξωτερικό. Όπως ξέρετε πρόκειται για μια δικασία που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ επίπονη και δύσκολη. Αυτά κυρία Πρόεδρε όσον αφορά τη γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Περνάω τώρα στους Σκιώδης. Πρώτη Σοφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Σικλούνα. Εξαιρετικά χρήσιμη πιστεύω η συζήτηση. Ακριβώς όπως είπατε κύριε Σικλούνα υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκίων των πολιτών και της καθημερινής τους εμπειρίας ε, λόγω της μεταφοράς των κειμένων που υιοθετούνται εδώ. Ε, αφορά το ζήτημα την ενία αγορά και από πολλές απόψεις είναι μια επιτυχία. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα δυσλειτουργίες και προβλήματα που αποτελούν το αντικείμενο της παρουσίας γνωμοδότησης. Επίσης, η οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς ε, που δεν έχει ως στόχο την υιοθέτηση απλά εκατοντάδων οδηγίων εναρμόνισης. Ε, στόχος είναι κυρίως ε, να παρακολουθούμε την καθημερινότητα των πολιτών μας και να βλέπουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί σε αυτή την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς. Ε, εγώ χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επιτροπός ε, Μπαρνιέ προσέχουν τη λειτουργία και παρακολουθούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση του συναδέλφου Ντουάρη είναι υψηλής ποιότητας και ότι καλύπτει τα ειδικότερα σημεία που αφορούν την το πεδίο εφαρμογή τη ΕΚΟΝ. Θα αναφέρω δύο-τρία που μου φαίνονται ουσιώδη σημασία. Μερικά από αυτά τα ανέφερε ήδη ο Εντουάρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια σημαντική πτυχή. Δηλαδή, η φραγμή, η φορολογική φραγμή στην καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ένα παράδειγμα που ανέφερε είναι η διπλή φορολόγηση. Εγώ συμφωνώ με την ανάλυση στην γνωμοδότησή του. Έχουμε ανοίξει τα σύνορα στους πολίτες. Πολλοί μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δουλειά τους, για τις συντάξεις τους, δεν είναι όλοι φορολογικοί εξόριστοι, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και τις διαφορετικές μορφές φορολογικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά οι κανόνες είναι υπερβολικά περίπλοκοι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αυτά τα φορολογικά θέματα. Πιστεύω, ωστόσο, ότι εδώ τίθεται θέμα ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εργαστεί και να παλέψει για αυτή τη φορολογική εναρμόνιση μίλησε για αυτό προηγουμένω και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει ο κύριος Σίκλουνα. Επίσης ο εισηγητής αναφέρεται στους φορείς αύξησης και στους φορείς ε, κοινοτομίας. Εμείς θέλουμε αυτή την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων ε, εργασίας, ειδικότερα και με τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Θέλω να σκεφτείτε επίσης, κύριε Σογητά, την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Γνωρίζετε ότι τα επενδυτικά ταμεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα για την οποία μιλήσαμε και χθες και προηγουμένως ε, συνάδει με τις ε, επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων. Πιστεύω ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερθούμε και σε αυτούς τους δύο φακέλους με τρόπο συνεκτικό και κοινό. Θα σας υπενθυμίσω, όπως είπε ο Επίτροπος ε, Μπαρνιέ, τον οποίο την ονομάζω πρόεδρο, είπε ότι 10% των επιχειρήσεων, 10% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 11 εκατομμύρια μισθωτοί οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι της ε, οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσθεθεί αυτό το κομμάτι στη γνωμοδότηση. Ωστόσο, συμφωνώ γενικά με τη γνωμοδότηση του εισηγητή, η οποία είναι εξαιρετική ποιότητας, και βάσει τη οποία θα μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τώρα τον κατάλογο σκηδιών και βλέπω ότι εγώ είμαι η μόνη σκηδιώδης, οπότε πρέπει να πω κάτι. Ε, ναι, το γνωρίζω Νικόλα, σε είδα. Ε, συμφωνώ Όσα έγραψατε, Εντουάρντ, είναι πολύ χρήσιμα και πολύ εύστοχα. Θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε όταν φτάσουμε σε φάση τροπολογιών, ε, ώστε να μην είσαι περιορισμένος όσον αφορά τα όρια πλήθους Αυτό που εγώ παρατηρώ, παρότι δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί αυτό στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας επιτροπής, θα πρέπει να μιλήσουμε για την κινητικότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων. Φαίνεται πολύ περίεργο να δημιουργούμε διάφορους κανόνες για τις συντάξεις και τις ασφάλειες ε, ζωής ε, και να πράττουμε κάτι τέτοιο διασυνοριακά όσο είναι δυνατόν, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να μεταφέρουμε μεγάλα χρηματικά ποσά από μια χώρα σε μια άλλη και ορισμένοι άνθρωποι όταν μετακομίζουν μπορεί να επιθυμούν να πράσουν κάτι τέτοιο. Συμφωνώ μαζί σου, υπάρχει ανάγκη ε, ευθυγράμμισης των δομών ΦΠΑ. Είναι από τα πιο συνήθι πράγματα, συνήθει καταστάσει που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανακτήσουν το ΦΠΑ από μια άλλη χώρα παρότι το δίκτυο Solvit ε, θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμο γι' αυτό. Επίσης κάτι άλλο που δεν αφορά απαραίτητα αυτήν εδώ την Επιτροπή, το ζήτημα των πινάκων συσχετισμού που γνωρίζουμε πάντα ότι της Επιτροπής της αρέσει να έχει ε, πίνακες συσχετισμών ε, και ξεκινάει με μια τέτοια φιλοδοξία στην νομοθετική διαδικασία, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να τους ε, να εφαρμόζονται παντού. Έχουμε θέσει το παράδειγμα σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Ένα single rule book βιβλίο νέων κανόνων ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτούς. Ε, πιστεύω ότι και σε άλλους τομείς πρέπει να ισχύει το ίδιο. Θέλω λοιπόν να ενθαρρύνω τους συναδέλφους από άλλες επιτροπές ίσως να το ζητήσουν λίγα και πιο στεναρά Είναι πιο δύσκολο φυσικά όταν ε, σε επίπεδο υλοποίηση, σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά ίσως ήδη σε επίπεδο, εκεί που δεν υπάρχει τέτοια περιφερειακή υλοποίηση, θα μπορούσαμε να τονίσουμε την απέτηση πινάκων συσχετισμών, ώστε να καταλάβουν όλοι ε, που βρίσκεται η νομοθεσία στη χώρα τους και στις άλλες ε, χώρες διότι διαφορετικά μιλάμε για ναρκοπαίδιο ακόμη και για όσους θέλουν να παράσχουν συμβουλές. Ε, είναι μια διαδικασία δαπανηρή και πρέπει κανείς να γνωρίζει πολλά ε, ώστε να μπορέσει να βγάλει άκρη. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια. Δεν βλέπω κάποιον από τους πρασινούς εδώ. Δάκα, έχεις το λόγο για το ECR. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω επικροτώντας αυτή την πρωτοβουλία. Μας υπενθυμίζει γιατί βρισκόμαστε εδώ η ενιαία αγορά είναι μια υπόσχεση που δεν έχει εκπληρωθεί σε την καθημερινή του ζωή. Οι πολίτε στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τι ανεπάρκειες όταν θέλουν να ασκήσουν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Μια πραγματικά ενιαία αγορά θα του παρέχει τη μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τόσο από τι χώρε του όσο και από το, όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Σε μια τέτοια αγορά τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα και οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν και να ζήσουν όπου θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση ο κύριος Σικλούνα δικαίως εστιάζεται στα ζητήματα στα οποία μπορεί να προσφέρει τη προστιθέμενη αξία η δική μας Επιτροπή στην Επιτροπή Εσωτερικής, Εσωτερικής Αγοράς ε, όπως η ανάγκη μείωση των, φραγμών, των φορολογικών φραγμών για τους διασυναριακούς εργαζόμενους και ε, εργοδότες, ε, τη μείωση της διπλής φορολόγησης και την πρόσβαση σε ενημέρωση για πολύπλοκα τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να κάνω μερικές άλλες προτάσεις όπως να αναφέρουμε ότι κύριο στόχο του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παρέχει κεφάλαιο στην πραγματική οικονομία. Ένα άλλο σημείο που θεωρώ σημαντικό είναι να ευαισθητοποιήσουμε του πολίτες ως προς τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η πρόταση του εισηγητή για τη ε, ε, χρηματοοικονομική ενημέρωση και εκπαίδευση. Επίσης, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της πλήρους δυναμικότητας της ενιαίας αγοράς με την πλήρη υλοποίησή της ε, της οδηγίας υπηρεσιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα θέσει τέλο στον κατακαιρματισμό τη αγορά και θα εξαλείψει του φραγμού στην ε, μετακίνηση υπηρεσιών, στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα. Εγώ ε, ε, εργαζόμουν στην προηγούμενη Επιτροπή Μπολκεστάν και θυμάμαι πως περιφρονούσαν αυτή την οδηγία και σήμερα βλέπω να αναζωογονείται. Ο ακόμη και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αναφέρεται σε αυτήν ως κύριο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Θέλω επίσης ο εισηγητής να εξετάσει να την αρχή της χώρας προέλευσης που έχει εγκαταλειφθεί από αυτή την οδηγία και να την υπανισάγει στο πλαίσιο μια διαδικασία βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών που το επιθυμούν. Δηλαδή κάποιο συνασπισμό ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ε, συγχαίρω τον κύριο Σεκλούνα με το σχέδιο γνωμοδότησης και προσβλέπω στην ε, πλήρη μας συνεργασία με τις τροπολογίες που θα υποβάλλω. Ευχαριστώ, Νικόλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας έκανε ό,τι μπορούσε τα θέματα που θίγει στη γνωμοδότηση είναι και υπαρκτά και σημαντικά. Όμως είναι παγιδευμένος στο πλαίσιο της έρευνας που έκανε η Επιτροπή και θα σας έλεγα και στον τίτλο που βάζει η Επιτροπή. Με αφορμή την έρευνα που έγινε για τα 20 χρόνια της ενιαίας αγοράς ήθελε να καταγράψει η Επιτροπή πώς αισθάνονται οι πολίτες και ποιες είναι οι κυριότερες ανησυχίες. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι οι κυριότερες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι αυτές που καταγράφει η Επιτροπή. Νομίζω ότι τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα τους απασχολούν πρώτον αν έχουν δουλειά, διότι γνωρίζετε τα νούμερα της ανεργίας, αν έχουν μισθό και πόσο θα περικοπεί. Τρίτο, αν υπάρχουν ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα ή εξανεμίστηκαν μέσα από αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά τους και τέτοια ερωτήματα. Πιθανόν να μου απαντήσετε ότι δεν είναι της δικής μας Επιτροπής. Αλλά για να είμαστε και αξιοπρεπής δεν μπορεί να μην, το δεις αυτό. Στην ίδια έρευνα άλλωστε, στην ίδια έρευνα η γνώμη των πολιτών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργασία και την κοινωνική πολιτική είναι αρνητική. Δηλαδή δεν προσδοκούν. Και επίσης το 62 έως 78% την ίδια έρευνα, για την ίδια έρευνα μιλάω, πιστεύει ότι δεν ενισχύεται η πρόσβασή τους στην εργασία και ότι δεν επιτυχάνεται η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή είναι η εικόνα και κατά τη γνώμη μου αυτές είναι οι κύριες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως φτιάχτηκε μια έκθεση, λέει 20 κύριες ανησυχίες και κατεγράφησαν ορισμένα, επαναλαμβάνω, υπαρκτά προβλήματα και τα προβλήματα που καταγράφει και ο εισηγητής μας είναι υπαρκτό, είναι σημαντικό, δεν το αρνούμε. Αλλά όμως δεν είναι η, βάση, η πραγματική βάση της όλης συζήτησης δεν είναι η πραγματική εικόνα της Ευρώπης. Δεν είναι οι πραγματικές κύριες, κύριες επαναλαμβάνω, ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Είναι πρόβλημα λοιπόν δυσλειτουργιών και προβλημάτων που καταγράφονται της εσωτερικής αγοράς ή είναι μια ευκαιρία, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το κάνουμε στη διάρκεια της γνωμοδότησης, να ξανασκεφτούμε η ενιαία εσωτερική αγορά είναι αυτός σκοπός. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε, να διορθώσουμε δυσλειτουργίες Κάποιο σκοπό πρέπει να έχει αυτό το πράγμα. Αν είναι η ευημερία των Ευρωπαίων, αν είναι να έχουν δικαιώματα, αν είναι για το μέλλον των παιδιών, πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικέ. Φυσικά η γνωμοδότηση δεν μπορεί να γράψει τέτοιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αρχική μου, η, η αρχική μας τοποθέτηση. Στο πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το ότι καταγράφονται εν τέλει σημαντικά πράγματα, με τροπολογίες να βοηθήσουμε να γραφτεί μια. Αλλά έχουμε αίσθηση μια καλή γνωμοδότηση. Αλλά έχουμε αίσθηση ότι δεν μιλάμε ούτε για τις κύριες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών, ούτε αυτά θα μπορέσουν να ανατρέψουν, να αλλάξουν την πολιτική και την κατάσταση ούτε ώστε πράγματι οι ανησυχίες των πολιτών να είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που ισχυρίστηκα εγώ και που βγαίνουν μάλλον από την έρευνα κομμάτια όμως τα οποία δεν αναφέρονται ας το πούμε ε, ως κύριες ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Edward. Ευχαριστώ, Edward. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλος το λόγο. Ε, ευχαριστώ τους και όσοι για τα σχόλιά τους. Τα σημείωσα όλα τα σχόλια, είναι πολύ χρήσιμα και περιμένω τροπολογίες ή να συναντάμε τους για ε, να συζητήσουμε. Και βεβαίως συμφωνώ με τον κύριο Χουντή. Στην έκθεσή μου όμως αναφέρονται οι ανησυχίες των πολιτών οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητα διασυνοριακά, να κάνουν ένα λογαριασμό σε μια άλλη χώρα. Κάποιο θέλει να κινηθεί, εργαζόμενο, εργοδότη. Με αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα μιλάμε εδώ. Δεν ε, μιλάμε γενικότερα για τις ανησυχίες του πολίτη στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω. Σωστά ανέφερε αυτά που ανέφερε. Και βεβαίως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα και ανησυχίες. Συμφωνώ μαζί του, αλλά το θέμα το δικό μου και το θέμα των σκιωδών εισηγητών είναι να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτά το οποίο αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 29 Μαρτίου προθέμενη κατάσταση τροπολογιών. Συζήτηση 25-26 Απριλίου ψηφοφορία 30, 31 Μαΐου, τον Ιούνιο η Επιτροπή και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια ψηφοφορία. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορούμε να περάσουμε λίγο ενωρίτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει στο επόμενο θέμα, το 15. Θέσφυση προγράμματος δράσης για τα τελωνία και τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φίσκους και την κατάργηση των αποφάσεων 1482 Παύλα 2007 και 624 2007. Πρόκειται για κοινό θέμα που επεξεργαζόμαστε με την ΙΜΚΟ αλλά ίσως κάποια στιγμή τα χωρίσουμε τα θέματα. Ήδη είχε μία συνάντηση από αυτού του θέματος η ΙΜΚΟ είμαστε ε, παρόντες, ήταν παρόν ο Παύλος Άλβα. Έχουμε εδώ μαζί μας την ΣΥΡΠΑ. Αλλά θα δώσουμε πρώτο το λόγο στον Θεοδόρ Στολογιάν που θα μας κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως βλέπετε πρόκειται για κοινή συνεδρίαση όπως προβλεπόταν μεταξύ της ΕΚΟΝ και της ΕΜΚΟ. Εδώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό βρισκόμαστε στο άρθρο 51 που προβλέπει κοινή συνεδρίαση, κοινή έκθεση και κοινή ψηφοφορία. Τι συμβαίνει όμως τώρα. Όπως ξέρετε η ΙΜΚΟ ήδη συνεδρίασε τη Δευτέρα και απεφάσισε και υποστήριξαν την ιδέα της δύο να χωρίσουμε την έκθεση για τα δύο προγράμματα, διότι το φίσκους αφορά πρώτα απ' όλα ε, τα τελωνία 2013 και το Φυσκάλι στην φορολογία 2013. Επίσης είπε η έκανε ότι θα πρέπει να χωριστούν αυτά τα δύο προγράμματα. Βάσει ποιων επιχειρημάτων. Θα σας τα παρουσιάσω συνοπτικά. Υπάρχουν δύο προγράμματα που λειτουργούν πολύ σωστά. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε υπήρξε η ενδιάμεση έκθεση αναθεώρησης. Έχουμε λοιπόν προγράμματα που λειτουργούν σωστά στους δύο αυτούς τομείς, τομείς που είναι διαφορετικής, οι στόχοι και η πολιτική που ακολουθείται επίσης είναι ε, ε, διαφορετική και φαίνεται ότι η υπάρχει μία κάποια συμφωνία κυρίως στον τομέα της φορολογίας. Αλλά υπάρχουν και ασυμφωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένω να επιβραδύνουν την πρόοδο που θα μπορούσε να επιτευχθεί στον τομέα των τελωνίων. Γι' αυτό, σύμφωνα με άτυπες πληροφορίες. Η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν τον διαχωρισμό αυτών των δύο προγραμμάτων, των δύο σκελών, αν θέλετε, του προγράμματος. Το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει αποφασίσει όσον αφορά το θέμα αυτό του διαχωρισμού. Επίσης, υπάρχει επιστολή του Επιτρόπου σε μέτα στην οποία εκφράζεται υπέρ του να έχουμε για τους δύο αυτούς τομείς, τα τελωνία και τη φορολογία, ένα ε, φάκελο, ένα πρόγραμμα αν θέλετε, δράσης. Διότι λέγει ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να φέρουν σε πέρας όλα τα θεσμικά όργανα είναι την απλοποίηση του πολιετές πλαισίου στον δημοσιονομικό κανονισμό. Υπάρχει λοιπόν ένα ενιαίο πρόγραμμα στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών κανονισμών και θα πρέπει να γίνει και τυποποίηση όλων των προγραμμάτων που αφορούν τους τομείς αυτούς όσον αφορά τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, την ε, ε, οικονομικό έλεγχο κτλ. Σε αυτή την επιστολή τονίζει επίσης ο Επίτροπος ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των φορολογικών συστημάτων και των τελωνιακών συστημάτων και η διαχωρισμός και η διαφοροποίηση μεταξύ τομέων και δράσεων καθώς και των κονδυλίων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, είναι ειδικοί στόχοι επιμέρους ο ένας για το τομέα της φορολογίας, επιμέρους ο άλλος για τα τελωνιακά και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό για αυτούς τους δύο τομείς, ο στόχος, ο αντικειμενικός τελικά είναι κοινός. Επίσης, υπάρχει εκ μέρου τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ε, γνωμοδότηση υπέρ του ενό ενιαίου προγράμματο δράση και θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτή την άτυπη έκθεση την οποία τις οποίες λάβαμε γνώση μετά τις συζητήσει που έγιναν στο Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία διάφορες χώρες μέλη πιστεύουν ότι το πρόγραμμα αυτό εισαγάγει νέους στόχους όπως ε, την εισαγωγή κάποιων νέων νόμων στους δύο αυτούς τομείς. Όσον αφορά την ουσία των προγράμματος δράσης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, αλλά εμείς θα πρέπει να βασίσουμε την εργασία μας στο άρθρο 51 προς το παρόν. Και όταν τελικά αποφασίσει το Συμβούλιο πώς θα προχωρήσει, αν θα τα χωρίσει τα δύο, το, πρόγραμμα αυτό σε δύο, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε εμείς τη δουλειά μας substance of the program. Όσον αφορά τώρα την ουσία, όπως σας είπα, υπάρχει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και ε, μελέτη αντικτύπων του φίσκους. Στον τομέα της φορολογίας Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ενώ το, το σκέλος τελωνία είναι θέμα αρμοδιότητας της ΣΥΜΚΟ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες στο δικό τους το κομμάτι των τελωνίων. Θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή, διότι έλαβε υπόψη την σύσταση τις συστάσεις που γίνονται στη μελέτη αντικτύπων και στην μεσοπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης. Και ποιος είναι ο κύριος στόχος. Η αποφυγή της απάτης, διασυνορικής απάτης, ε, αποφυγής, φορολογίας, προστασία των φορολογουμένων, έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν τους τομείς αυτές και την ανάπτυξη ενό ε, ασφαλούς δικτύου ανταλλαγή προφορίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι συστάσεις ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή για την συγκρότηση του προγράμματος και συνεργασία με τρίτες χώρες και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Εκτός από αυτά τα οποία ξέραμε για το ΦΠΑ, για τους έμεσους φόρους κτλ. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να καλύψει και νέους στόχους όπως αμοιαία σύνδρομη για την ανάκαμψη πόσο που το τάξ, τους φόρους, ενεργειακά κτλ. Όσον αφορά τη συμμετοχή. Υπάρχει μια κοινοτομία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδεχόμενες υποψήφιες χώρες και προτείνει νέους εταίρους για αυτό το πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ε, χώρες χώρες-εταίρες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Γειτονίας εφόσον οι χώρες αυτές έχουν προσαρμόσει ε, παρκώς τα ε, κανονισμούς που τους διέπλουν και τα θεσμικά τους όργανα ώστε να μπορέσουν σύμφωνα με τα δικά μας δικές μας επιθυμίες και δεδομένα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όσον αφορά τις επιλέξιμες δράσεις, προτείνει η Επιτροπή να διατηρήσουμε τις ίδιες δομές. Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, κοινέ δράσεις Δηλαδή ανταλλαγή πρακτικών, ε, γνώσεων, τεχνογνωσίες, δημιουργία ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφόρησης, δραστηριότητες κατάρτισης και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως, το πρόγραμμα αυτό είναι στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και τα προγράμματα τα παρελθόντα και αυτό το πρόγραμμα είναι προγράμματα τα οποία εφαρμόζει η Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη και η διαχείρισή τους έχει αναλυφθεί από την Κομισιό όσον αφορά τα κονδύλια, τον προϋπολογισμό. Υπάρχει συνολικό ποσό. Έχουμε 777,6 εκατομμύρια ευρώ. 554 πάνε στον τομέα των τελωνίων, δηλαδή το 70%. Και για την τομέα της φορολογίας 332,2 δηλαδή 30%. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε για τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό είναι ότι βεβαίως σε κανέναν δεν αρέσει το μέσο φορολογίας. Φαίνεται και αυτή είναι η πρώτη μου, ε, να το πω, αξιολόγηση και παρατήρηση Υπάρχουν ε, ελλειπή κονδύλια για αυτό το τομέα. Στο προηγούμενα προγράμματα, αν λάβουμε υπόψη της κρίσης της Επιτροπής για το πολιετές πλαίσιο, λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς κάποιο έτος και κάνοντας πολλαπλησιασμούς που χρειάζεται, φαίνεται ότι στον τομέα αυτό δεν πηγαίνουν καθόλου κονδύλια ένα όλα στον άλλο. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι κάποιοι πολύπλογοι υπολογισμοί. Και στο προηγούμενο πρόγραμμα τα κονδύλια για τα τελωνία ήταν το 67% ενώ τώρα υπάρχει μια μικρή αύξηση και είναι το 70% και το ΜΕΑΣ Συγγνώμη, αυτά είναι τα τελωνία. Ενώ προηγουμένω είχαμε για την φορολογία 33% και τώρα κατεβήκαμε στο 30%. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, ο τομέας της φορολογίας εμφανίζεται πιο φτωχός είναι ο φτωχό συγγενή αυτού του προπολογισμού. Αν δούμε λοιπόν τη δομή του προπολογισμού αυτού, το IT, η ανάπτυξη, η συντήρηση σημαίνει 81% για τα τελωνία και το υπόλοιπο για τα φορολογικά. Τα περισσότερα χρήματα λοιπόν δίνονται για το IT. Για τον, τον τομέα των πληροφοριών. Για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών όπως λέγεται, όπως ονομάζεται. Στον τομέα των τελωνίων υπάρχει και επίσης σημαντικό αύξηση που προβλέπεται για κοινέ δράσεις, σεμινάρια, συζητήσεις, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστες πρακτικές και στον τομέα της φορολογίας μόνο αύξηση για κατάρτιση. Αύξηση των κονδυλίων για κατάρτιση. Αυτά σας λέω σε πρώτη φάση και θα με ενδιέφερε να έχω τις δικές σας απόψεις, πρώτα απ' όλα τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Um, λοιπόν, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Εγώ όσον αφορά την συγχώνευση. Συμφωνώ με το πρόγραμμα Φίσκος και καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να μειώσει τα προγράμματα, τον αριθμό των προγραμμάτων τουλάχιστον, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει χωρίς συνοχή. Και βεβαίως τα προγράμματα των τελωνίων και των φυσκάλης δεν έχουν αρκετή συνοχή αν θέλετε έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει συγχώνευση. Μέχρι τώρα τα προγράμματα αυτά έχουν λειτουργήσει από μόνοι τους ξεχωριστά πάρα πολύ ικανοποιητικά. Όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος, βεβαίως και είμαι υπέρ του να βελτιώσουμε την ανταλλαγή των πληροφοριών, τις ε, βέλτιστες πρακτικές και βεβαίως να ενισχύσουμε και τα τεχνικά μέσα, την πληροφορική, αλλά και τους, ε, τα δίκτυα των ε, συμμετεχόντων. Πρέπει να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Καθότι σε μια εποχή οικονομικής κρίσης αυτό είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και την Σύρβα Πιτικάινεν, μέσω της ΙΜΚΟ, και μετά θα επανέλθουμε στους κοιότης. Ευχαριστώ. Ναι, πολλές φορές έχουμε πολλές ιδιότητες. Είμαι μέλος της ΣΥΜΚΟ, αντιπρόεδρος, μόλις εξελέγην και η συγγήτρια, μάλλον ο εισηγητής ο κύριος Μπαλτασά δεν μπορεί να είναι παρόν. Γι' αυτό και εκπροσωπώ εδώ τη θέση της ε, ΙΜΚΟ. Σύντομα βέβαια, ο κύριος Στολόγιαν παρουσίασε τα περισσότερα στοιχεία και ήθελα να σας πω ότι όταν Ακούσαμε τον διευθυντή της Taxud. Όντως, ε, ο κύριος στόχος είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η πιο αποτελεσματική δράση. Και βεβαίως, ε, ειλικρινά, όταν ακούσαμε αυτές ε, τις ιδέες, Όντως ε, το να υπάρξει συγχώνευση, συντονισμός και συνοχή είναι κάτι το πάρα πολύ λογικό. Οι στόχοι αυτοί είναι καθοριστικοί για να υπάρξει πραγματικά καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ΙΜΚΟ λοιπόν καταρχήν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μελέτη αντικτύπου σε δύο διαφορετικά τμήματα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε κατανοήσει ακριβώς τι θα σημάνει το να συγχωνευτούν αυτά τα δύο στοιχεία. Δεύτερον, αυτά τα δύο ξεχωριστά προγράμματα είναι πάρα πολύ επιτυχή ξεχωριστά από μόνα τους. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, λόγος ή ε, απόδειξη ότι αυτά τα δύο προγράμματα θα λειτουργήσουν καλύτερα από κοινού, αν συγχωνευτούν. Δεν βλέπω δηλαδή ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία ή το απτό αποτέλεσμα αν συγχωνευτεί το ένα πρόγραμμα με το άλλο. Η Επιτροπή λέει απλοποίηση, ε, απλούστευση κτλ και βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε καθυστέρηση όσον αφορά τα τελωνιακά προγράμματα και γι' αυτό και η αντίδραση της ΙΜΚΟ ήταν μάλλον αρνητική σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Βλέπω ότι ο, ο, ε, ο του Άλντι δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, οπότε παίζω δύο ρόλους, ε, και το δικό μου και το δικό του. Μου έχει δώσει ένα σημείο θα είμαι αρκετά σύντομη, λέγοντας ότι ο Κλίντα ε, υποστηρίζει την ενσωμάτωση των δύο προγραμμάτων για διάφορους λόγους. Ε, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη αναλυθεί και διερευνηθεί η, το, η αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, για παράδειγμα, για το τελωνιακό πρόγραμμα και οι πτυχές της ε, εσωτερικής αγοράς ε, για τα τελωνία και στη συνέχεια το γεγονός ότι η φορολογία υλοποιείται με τρόπο προσανατολισμένο στα κράτη-μέλη. Η ερώτηση που έγινε από τον εισηγητή αφορά, είναι πολύ σημαντική και αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και παρόμοια φαινόμενα, θα πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται και να είμαστε βέβαιοι ότι ο προπολογισμό κατανέμεται σωστά και αυτό θα μας βοηθήσει. Ο Δ. Κλίντ είναι επίσης πεπισμένος ότι λαμβάνει κανείς, ότι επιτυχάνεται μείωση με τη συγχώνευση δύο προγραμμάτων ε, αλλά όχι με τη συγχώνευση των δύο προγραμμάτων, αλλά με, τις, με επιμέρους μειώσει σε καθένα από τα προγράμματα, διότι αλλιώ είναι πολύ περίεργο ο χειρισμό και των δύο προγραμμάτων μαζί. Βλέπω ότι είναι περίεργο και εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι δύσκολο για το μέλη του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε δύο συνεδριάσεις αντί για, σε... αντί για μία. Σίγουρα αυτό δεν απλοποιεί τα πράγματα εντός του Κοινοβουλίου σε καμία περίπτωση. Η κοινή μας άποψη λοιπόν από το Άλντι μαζί με το ΑΛΔ ότι θέλουμε να είναι ξεχωριστά. Περνάω στον επόμενο σκιώδη. Φιλίπ, είσαι εδώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι όταν εξαναγκάζει κανείς ανθρώπους να συμμετέχουν σε δύο συνεδριάσεις, τους δίνει κανείς μια δικαιολογία για να μην βρεθεί σε καμία συνεδρίαση. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και εξοικονόμηση πόρων, παρότι δεν νομίζω ότι έτσι συμβαίνει γιατί βλέποντας ε, το πλήθος ε, ε, προσωπικού και διερμηνέων που βρίσκονται εδώ για έξι μόνο μέλη του Κοινοβουλίου. Οι διερμηνείς είναι εδώ και για το web streaming. Φυσικά είμαι σίγουρος ότι έχουμε και πολλούς θεατές αυτή τη στιγμή τέτοια ώρα της ημέρας και για ένα τόσο συναρπαστικό ζήτημα. ούτως ή άλλως αυτό μας αποτελεί μια ένδειξη του πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε δαπάνε στο κοινοβούλιο. Δεν έχω κάποια άποψη για το αν πρέπει να τα συγχωνεύσουμε ή όχι. Ε, ξέρω ότι εσείς φιλελεύθεροι θα επιλέξετε οποιαδήποτε λογική επιλογή για εξοικονόμηση δαπανών. Ε, αν βλέπετε λοιπόν μια ευκαιρία, δεν τη χάνετε είμαι βέβαιος ε, και εγώ θα το δεχτώ την κρίση ανθρώπων πιο έμπρον από εμένα. Τώρα, επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτός είναι ένας τομέας φορολόγησης όπου έχουμε συναπόφαση. Αυτό το επικροτώ. Θέλω αυτό να αξιοποιηθεί για ολόκληρο το κονδύλιο θα ήθελα να διερευνήσουμε κατά πόσο όταν ξεκινάμε και μιλάμε για ένα μέσο συνεργασία μεταξύ φορολογικών διοικήσεων, μήπω θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να εισαγάγουμε μέτρα όπω ε, για παράδειγμα γιατί να μην ενεργοποιήσουμε ή εξαναγκάσουμε τι φορολογικέ διοικησει, να μοιράζονται δεδομένα σε σχέση με τι ε, φορολογικέ αποφάσει για επιμέρου εταιρείε. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, οι εφορέ του Λουξεμβούργου λαμβάνουν αποφάσεις ε, φορολογικέ ε, στο Βέλγιο επίση χωρίς να ξέρει ο άλλο. Ε, και έτσι λοιπόν έχουμε διπλή, τριπλή, τετραπλή μη φορολόγηση και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο στην παρούσα το μόνο που θέλω να πω ανεξαρτήτως του αν θα κρατήσουμε τα προγράμματα ξεχωριστά ή θα τα συγχωνεύσουμε. Θα ήθελα να το αξιοποιήσει όλο αυτό το κοινοβούλιο στο μέγιστο βαθμό ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ε, δημόσιο εχθρό ουσιαστικά που είναι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Αυτές οι φορολογικές αποφάσεις λοιπόν είναι κάτι που με απασχολούν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήβο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώντας ε, θα συνεχίσω με την ίδια σκέψη κοιτώντας γύρω μου Φαίνεται σαν να είμαστε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Και η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι, κυρία Πρόεδρε, εσείς βρίσκεστε ακόμη εδώ και έχετε τόσο μεγάλη υπομονή με όλους μας. Ε, δεύτερον, εκτιμώ την παρουσία όλων των διερμηνέων που κάθονται τριγύρω μας και κάνουν τη δουλειά τους ε, άριστα. Και έχω και μερικές παρατηρήσεις τώρα για τις παρατηρήσεις του κυρίου Στόλογιάν. Θα προσπαθήσω να βγάλω άκρη από τις χάουδες δικές μου σημειώσεις. Ε, η πρώτη, ειλικρινά, προσπάθησα να βρω πιθανές πήγες για το φίσκους, όπως ε, αναφέρατε εσείς κύριε Στολογιάν. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να βρω τις απαραίτητες λεπτομέρειες. μαζί με όλους εσάς πιστεύω είμαι σκεπτικός όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο μου σημείο, εφόσον έχω καταλάβει καλά, το πρόγραμμα φίσκους θα πρέπει να είναι κάτι σαν διάδοχος του Customs 2013 και του Fiscalis 2013 αλλά και τα δύο προγράμματα στο εσωτερικό τους είναι αρκετά διαφορετικά από άψη περιεχομένου και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Το customs ε, με ένα πιο ενωσιακό ή στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και η φορολόγηση σε, πιο, σε πλαίσιο αρμοδιοτήτων κρατών μελών. Από αυτή την άποψη κατανοώ ή θα μπορούσα να καταλάβω, θα μπορούσα να δείξω κάποια κατανόηση γιατί ο προϋπολογισμός είναι αναλογικά διαφορετικός. Δύο τρίτα στα ε, τελωνία και ένα τρίτο για τη φορολόγηση. Σεβόμενος φυσικά τις αρμοδιότητες μου φαίνεται κατανοητό το να δώσουμε 80% στα ε, τελωνία και το 20% στη φορολόγηση. Το καταλαβαίνω. Πιστέψτε με αν θέλετε, αλλά πραγματικά, ακόμη και μετά τις δικές σας παρατηρήσεις, προς το παρόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και τα δύο προγράμματα δεν θα μπορούσαν να συνεπάρχουν παράλληλα. Για ποιο λόγο το ένα πρόγραμμα θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο κατ' εμέ είναι αμφισβητήσιμο. Προς το παρόν δυσκολεύομαι να καταλάβω ποιο θα ήταν το σημαντικό όφελος, ίσως εξοικονόμηση χρημάτων όπως ακούσαμε, το οποίο εγώ θα εκτιμούσα ιδιαίτερα, αλλά δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Αναμένω ότι να συνεργαστούμε κύριε Στολογιάν, και θα δούμε σύντομα η λίγο αργότερα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκο Χουντή ήταν σκιώδη του Σγκούε. Δεν ξέρω, Γιώργη, αν θε να πει κάτι. Ενώ ο Νίκο είναι απασχολημένο. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στο ΑΦΕΤ, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Συνεπώ δεν μπορούσε να είναι μαζί μα και δεν έχω ετοιμαστεί εγώ για το θέμα. συγγνώμη. Ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να ζητάει το λόγο από τα μέλη. Φυσικά ακούσαμε ήδη τον Επιτροπό γιατί το αναφέραμε στην ανταλλαγή απόψεών μας με τον Επιτροπό νωρίτερα αυτή τη βδομάδα. Και ορισμένοι έχουν μάθει από άλλα μέλη της Επιτροπής. Κυρία Μπόλς, μήπως ε, θα μπορούσε να μας ενημερώσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου αν βρίσκεται εδώ ε, για αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον από την Προεδρία εδώ. Και οι επιμέρους αντιπροσωπείες δεν νομίζω ότι μπορούν να αναλάβουν τέτοια ευθύνη. Δεν υπάρχει κανείς από την Προεδρία, όχι. Ζήτω συγγνώμη λοιπόν, είναι αδύνατον. Δεν βρίσκεται κανείς εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Βρισκόμαστε σε, σε μια αφετηρία. Συμφωνώ τα με την ιδέα της επανεστίασης του προγράμματος. Στην πραγματικότητα η πρόταση της Επιτροπής υπογραμμίζει την επανεστίαση των στόχων για την καταπολέμηση της απάτης διασυνοριακά, της φοροδιαφυγής και ίσως θα έπρεπε στις, να, στις τροπολογίες μας ε, να επισημάνουμε περισσότερο την ιδέα αυτή στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα. Ναι, συμφωνώ. Τη δομή και του προϋπολογισμού. Η δομή του προϋπολογισμού φυσικά εστιάζεται κατά 80% ε, για τα τελωνία και τα IT ενώ 20% για τον τομέα της φορολόγησης ε, και για τα IT. Ε, αυτό συνέβη και με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζω καλά αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο με την Κομισιόν αυτό το ζήτημα είναι γιατί σύμφωνα με το δικό μου υπολογισμό ο προπολογισμό για, τα... για το τελωνιακό σύστημα αυξάνεται ενώ ο προπολογισμό για το φορολογικό τομέα παραμένει ίδιος σχεδόν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διασαφηνίσουμε και να, θα πρέπει να έχουμε σαφή επιχειρήματα εκ μέρους της Κομισιόν. Το πρόβλημα τώρα, κυρία Μπόλς, αν ε, πρόκειται εδώ να συζητήσουμε μόνο το αν θα συζητήσουμε μόνο εδώ το φορολογικό κομμάτι οι συναδελφοί μου από την εικόνα θα σκέφτονται ότι είναι καλή δεν μπορεί να μας απαγορέψει να κάνουμε τροπολογίες, να ε, συζητήσουμε και το τελωνιακό κομμάτι του προγράμματος. Αλλά ουσιαστικά η στίωση των συναδέλφων μου στην όπως πιστεύω εγώ, θα είναι να εστιαστούμε στο φορολογικό κομμάτι και οι συνάδελφοι της ΙΜΚΟ θα μπορέσουν να συνεισφέρουν όσον αφορά τα τελωνία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μια άλλη πτυχή της παρουσίασης της Κομισιόν η οποία αφορά το, το κομμάτι της φορολόγησης στο κοινό πρόγραμμα. Είπατε καθαρά, ο κύριος λάμπερτο, μίλησε για συναπόφαση επειδή το Κοινοβούλιο σήμερα βρίσκεται σε στάδιο συναπόφασης για αυτό το φορολογικό πρόγραμμα. Για ποιο λόγο, διότι αυτό το πρόγραμμα αντιμετωπίζεται από την Κομισιόν ως ε, τρόπος βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, Υπάρχουν περισσότερα επιχειρήματα για την τήρηση της επικουρικότητας. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή παίζει σαφή ρόλο στη διαχείριση του προγράμματος αυτού για το φορολογικό τομέα. Δεν έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε ότι αν υπάρχει φορολογικό ζήτημα όπου τα κράτη-μέλη είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να λαμβάνουν αποφάσεις και να συμφωνούν για ζητήματα φορολογικά ομόφωνα με, με ψήφους ομοφωνίας. Ε, τώρα συζητάμε ένα πρόγραμμα το οποίο σαφώς εστιάζεται στην υποστήριξη της σωστή λειτουργία του, των φορολογικών συστημάτων μέσω της συνεργασία, μέσω αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και επίσης ε, για την οικοδόμηση, την ανάπτυξη την ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών. Ουσιαστικά μέσα στο πρόγραμμα αναφέρεται πολύ καθαρά. Στην εισαγωγή του προγράμματος αναφέρεται καθαρά ότι έχουμε ένα πρόβλημα ακόμη λόγω των διαφορετικών πληροφορικών συστημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη, τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τάση. Αύξηση των πληροφορικών συστημάτων, μάλιστα. Ε, κύριε Μπόλζη, η Κομισιόν επίσης επέκρινε έκρινε μάλλον την ενδεχόμενο εξωτερήκευση αυτού του προγράμματος. Αυτό σημαίνει δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό υλοποίηση αυτού του προγράμματος και το συμπέρασμα είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστάται. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση προκύπτει ότι τα προγράμματα όχι μόνο υλοποιήθηκαν πολύ καλά όσον αφορά τα αποτελέσματά τους αλλά και όσον αφορά τη διαχείρισή τους απόψη προβλημάτων και ούτω καθεξής. Τώρα όμως έχουμε ένα νέο οργανισμό για την πληροφορική που έχει ιδρυθεί στην Εστονία, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Διότι αυτός ο οργανισμός, νέος ευρωπαϊκός οργανισμός πληροφορικής, ίσως να ψάχνει να βρει δουλειά σε λίγο. Και αν αυτός ο οργανισμός αρχίσει να ψάχνει για δουλειά, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ένα, ένα καινούριο πρόβλημα. Θα πρέπει να αποφασίσει ποιο κομμάτι αυτή τη πληροφορική που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού εδώ του προπολογισμού θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιο κομμάτι θα μεταβιβαστεί σε αυτόν τον νεοσύστατο οργανισμό στην Εστονία. Μόλις έμαθα για τη δημιουργία αυτού του οργανισμού στην Εστονία σήμερα και οπότε θα σκεφτούμε και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, καλός τρόπος εξοικονόμησης λοιπόν δημιουργία ενός οργανισμού. Όσον αφορά την ερώτησή σου, Θεόντορ, για το πώς θα προχωρήσουμε, αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό το άρθρο 51, διότι η πρόταση Ουσιαστικά ήταν διαχωρισμό 50%-50% μεταξύ των δύο επιτροπών. Έτσι λοιπόν υποχρεούμαστε να συνεδριάζουμε μαζί. Αλλά όσον αφορά τα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούμε, φυσικά εμεί θα επικεντρωθούμε ε, στις στι αντίστοιχε των επιτροπών μας. Φυσικά, αν καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τα δύο ζητήματα, τότε θα έχουμε δύο ξεχωριστές εκθέσεις. Και τέλος, ε, αν εξακολουθήσουμε να συνεδριάζουμε μαζί, τότε όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας τότε όλοι θα ψηφίσουμε για όλες τις τροπολογίες. Εάν λοιπόν έχουμε προτείνει κάτι το οποίο αφορά τα τελωνία, φυσικά το προσωπικό της ΕΜΚΟ θα το, εξετάσει και αυτοί, θα το εξετάσουν και αυτοί. Αλλά όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και στις πολιτικές μας ομάδες για συμβιβασμούς και κοινέ λύσεις της ψηφοφορίας. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την εμπειρογνωμοσύνη της εκάστοτε επιτροπής και σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε λογικά έτσι ακριβώς όπως κάνουμε σε περίπτωση ενισχυμένης συνεργασίας. Το θέμα λοιπόν παραμένει ανοιχτό το κατά πόσο θα συνεδριάζουμε μαζί ή αν ε, χάρη στην ομόφωνη θέση των δύο επιτροπών δεν επιθυμήσουμε να συγχωνεύσουμε αυτά τα δύο ενώ θα μπορούσαμε. Ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος τώρα είναι να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την εκθέσή σα μέχρι τις 25 Απριλίου. Τροπολογίες για τις 7 Μαΐου, συζήτηση στι 30 Μαΐου και ψηφοφορία στι 7 Ιουνίου. Αλλά όλα αυτά παραμένουν ρευστά. Θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Μπορεί να γίνει ίσως πιο αργά για να το πω διπλωματικά. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη για την παρουσία τους. Δεν έχουμε κανένα θέμα στα διάφορα, οπότε μπορούμε να φύγουμε, γιατί και εγώ πρέπει να πάρω το αεροπλάνο για την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.